So, good morning, ladies and gentlemen. Uh, uh, ναι, ο κύριος Λόπες Αγγιάρο, ο πρόεδρος μας, ε, είναι σε συνεδρίαση. Ε, άλλος αντιπρόεδρος δεν είναι ελεύθερος και έτσι μου ζητήθηκε να αναλάβω εγώ την καθοδήγηση της ε, συνεδριάσεως σήμερα. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα γνωρίζετε ίσως ότι η Επιτροπή των Νομικών Υποθέσεων συντάσσει έκθεση Δίας Πρωτοβουλίας όπου καταγράφει τις εξελίξεις ως προς τις κατεξουσιοδότηση πράξεις και τις εκτελεστικές πράξεις, κάτι το οποίο έχει πολύ μεγάλη σημασία για τις εργασίες της δικές μας βέβαια. Δυστυχώς το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν διάκυνται θετικά, πολλές φορές μάλιστα είναι κατά των κατεξουσιοδότησης πράξεων. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε εμείς είναι να μιλήσουμε για τις ε, εκτελεστικές πράξεις. Σήμερα θα ακούσουμε την κυρία Πρίσκοβα Μπένοβα, την συγκητρία μας, η οποία θα μας παρουσιάσει το σχέδιο γνωμοδότησης της. Στο θέμα αυτό και στη συνέχεια θα δώσω το λόγο στους λοιπούς συναδέλφους που θέλουν ε, να παρέμβουν. Έχετε το λόγο, Μόνικα. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι. Όπως πήγε η κυρία Πρόεδρος. Πρόκειται για μια έκθεση μεγάλης ε, σημασίας σε πολιτικούς όρους, γιατί έχει ιδιαίτερα εφαρμογή στο σύστημα PNR, δηλαδή την ε, συλλογή και διατήρηση δεδομένων ε, επιβατών, κάτι το οποίο θα κριθεί εάν θα ε, υλοποιηθεί με βάση το, τις εκτελεστικές ή τις ε, ε κατεξουσιοδότηση Τρία χρόνια μετά τη Λισαβόνα, αποφάσεις οι οποίες έχουν μεγάλη πολιτική σημασία και αντίκτυπο δεν, δεν ε, αφήνουν περιθώριο για τοποθέτηση στους πολιτικούς. Πρέπει λοιπόν η Νομική Επιτροπή να παρέμβει για να εντοπίσει τους τομείς αυτούς με τα άρθρα 90-91 που ορίζουν τον τρόπο λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις ε, κα... Ε, κατεξουδότης συμπράξης, τη διαδικασία. της Επιτροπολογίας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λοιπόν ε, όταν πρόκειται για τέτοια βασικά θέματα θα πρέπει να αποφασίζει μαζί με το Συμβούλιο και την Επιτροπή ουσιαστικά πολιτικά ζητήματα και δευτερεύουσα σημασίας θέματα που δεν έχουν ουσιώδη βαρύτητα αλλά πρέπει να αντιμετωπιστούν εφόσον έχουν καλυφθεί τα πολιτικά, οι πολιτικές, τα πολιτικές μέρημνες ε, μπορούν να επιληθούν με την καταδεξιδότηση πράξη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, σε μεταγενέστερο στάδιο. Κάθε της πράξη, ωστόσο, επαληθεύεται από το συνομοθέτη. Το Συμβούλιο δηλαδή και το Κοινοβούλιο έχει το δικαίωμα της άρνηση κυρίας ε, στην περίπτωση όπου διαπιστώνει ε, υπέρβαση των ορίων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Άλλη περίπτωση είναι οι εκτελεστικές πράξεις που συνήθως υιοθετεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και προτείνονται για ε, επαλήθευση από τα κράτη-μέλη. Αυτές όμως μπορούν να υλοποιηθούν μόνο, να χρησιμοποιηθούν μόνο όπου υπάρχει ανάγκη για την εφαρμογή ομοιόμορφων όρων εφαρμογής ενός νομοθετήματο. Και τρία είναι τα βασικά και τα κρίσιμα σημεία στα οποία περιστρέφεται η γνωμοδότησή μας. Πρώτα απ' όλα έχουμε τον τρίτο πυλώνα, μια σειρά από ζητήματα που δεν έχουν αναθεωρηθεί από τη συνθήκη της Λισαβόνας, ε, νομοθετήματα τα οποία ε, δεν ανήκουν στο ανώτερο επίπεδο ιεράρχησης της ε, σειράς που έχει ορίσει η συνθήκη της Λισαβόνας, σειρά νομοθετημάτων για τα οποία δεν έχει αρμοδιότητα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ιδιαίτερα όσον αφορά τις κατεξουδότητες πράξεις και θα πρέπει ιδιαίτερα να δοθεί έμφαση στα ζητήματα του τρίτου πυλώνα. Καλούμε λοιπόν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταθέσει προτάσεις για να ε, ευθυγραμμίσει τις πράξεις αυτές με τους όρους τη συνθήκη τη Λισαβόνα. Ξέρουμε ότι δεν είναι ευχερέ το έργο, γιατί κάθε νομοθέτημα θα πρέπει ανεξάρτητα από τα υπόλοιπα και βάσει με, τη, με τα ιδιαίτερά του χαρακτηριστικά να αξιολογηθεί. και επίσης πολύ συχνά βλέπουμε αντίσταση από το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως προς τις δικές μας τροπολογίες κατά εξουσιοδότηση πράξη, ακόμη και όταν πληρούνται τα, οι προϋποθέσεις για μια κατεξουδότηση πράξη. Το πεδίο λοιπόν είναι πολύ ευρύ, αλλά πολύ συχνά το Συμβούλιο και η Επιτροπή αντιδρούν, αντιτίθενται σε τέτοιες πράξεις γιατί δεν θέλουν ε, να συμμετέχει το Κοινοβούλιο και να επιβλέπει και τις κατεξουδότηση σε αυτές πράξεις. Προτιμούν δηλαδή να καλύπτονται όλες τις λεπτομέρειες, να ρυθμίζονται όλα τα ζητήματα από τις εκτελεστικές πράξεις όπου μόνο ρόλο παρατηρητή μπορεί να έχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και έτσι ε, κάποιοι συνάδελφοι που έχουν αναλάβει εκθέσεις για θέματα συναπόφασης θα ήταν σκόπιμο και τους καλούμε να ε, συνεργαστούν μαζί μας και να συνομιλήσουν με το Συμβούλιο και την Επιτροπή και για τα θέματα των κατεξοδότησης πράξεων. Ένα τρίτο ζήτημα το οποίο θα ήθελα επίσης να αναφέρω ήταν ε, στην τρίτη αιτιολογική πρόταση το η αναφορά στο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο όπου η δέσκευση των Προέδρων, ξέρουμε, έχει ε, τοποθετηθεί με μια γνωμοδότηση λέγοντας ότι θα πρέπει να ε, εργαζόμαστε με τις εν πράξεις. Το Συμβούλιο και η Επιτροπή όμως ε, τάσσονται κατά της ρύθμισης τέτοιων προγραμμάτων πολιτών δημοσιονομικών προγραμμάτων μέσω εν συμπράξεων. Εμείς όμως ως Κοινοβούλιο είμαστε υπόλογοι εναντί των ψηφοφόρων μας, εναντί του εκλογικού σώματος και τον τρόπο με τον οποίο δαπανώνται τα ευρωπαϊκά κονδύλια, για τις προτεραιότητες που ορίζονται, εφόσον έχουν δηλαδή προσδοριστεί μέσα από τον τριμερή διάλογο, πρέπει να γίνεται και αντίστοιχα η δαπάνη, η εκτέλεση της δαπάνης. Αυτό σημαίνει εκτελεστικές πράξεις και για τα δημοσιονομικά προγράμματα, ετήσια ή πολυετή, τα οποία θα ε, υιοθετούνται με βάση τα δημοσιονομικά προγράμματα. Αυτά είναι τα σημεία στα οποία θα ήθελα να αναφερθώ στην γνωμοδότησή μου. Το σχέδιο εγγράφου εργασίας του εισηγητή του, της Επιτροπής των Νομικών Υποθέσεων πριν, πριν μερικές μέρες μόνο δημοσιεύτηκε. Εγώ παρακολουθώ φυσικά τις εργασίες της νομικής και το έγγραφο εργασία θα το μελετήσω πολύ προσεκτικά και βεβαίω το σχέδιο εκθέσεως Επιτροπής ώστε να κρίνω αν χρειαστούν επιπλέον ε, παρατηρήσεις στο σχέδιο γνωμοδότησής μας και τροποποίησης. Ενδεχομένως να καταθέσω τροπολογίες. Ε, Πάντω τώρα περιμένω να ακούσω του συναδέλφου και ο ή λοιπού, λοιπά μέλη τη Επιτροπής για τι πράξει αυτέ και βέβαια μέσα στι επόμενε εβδομάδε θα μα απασχολήσει το θέμα αυτό, Στι επόμενε μέρε θα το ξαναδούμε. Πρέπει να συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια γιατί πρόκειται για θέματα πολύ μεγάλη σημασία για την Επιτροπή μας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Και τώρα να δώσω το λόγο σε όποιον επιθυμεί, έτσι ώστε να λάβει χώρα συζήτηση, αν βεβαίως κάποιος θέλει να εκφράσει τη δική του ή δική της γνώμη. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Λέει ο κύριος Μέλο. Μια ερώτηση θέλω να υποβάλω, η οποία αφορά τον ε, μηχανισμό στον οποίο αναφέρθηκε η συνάδελφος στο τέλος της παρέμβασής της. Ξαναρχίζω λοιπόν, γιατί μιλούσα λίγο μακριά από το μικρόφωνο. Ε, να σας πω λοιπόν ότι έφτασα την ώρα που ολοκλήρωνε η συγκήτρια ε, την παρέμβασή της. Γι' αυτό δεν ξέρω εάν αναφέρθηκε στο θέμα περί του οποίου θα υποβάλω ε, ερώτηση. Αναφέρομαι στην αποτελεσματικότητα ή όχι ε, του μηχανισμού ελέγχου που προβλέπεται από, το, από τον 182 ε, του 2011, βάσει του οποίου ε, πρέπει το Συμβούλιο και η Κομισιόν να διαβουλεύονται ε, τακτικά με μια επιτροπή η οποία αποτελείται από διάφορα μέλη, εκπροσώπους κρατών, κοινοβουλίων κτλ. Θα ήθελα λοιπόν ε, να μου πείτε τι μπορούμε να κάνουμε στα πλαίσια της δικής σας γνωμοδότησης έτσι ώστε να βεβαιωθούμε ότι στο μέλλον δεν θα αμφισβητήσει η Κομισιόν ε, την συζήτηση για τις κατεξουσιοδότηση πράξεις. Ε, οι εκτελεστικές πράξεις μπορούν να μπλοκαριστούν από το Κοινοβούλιο στις ε, κατεξουσιοδότηση πράξης έχει δυνατότητα το Κοινοβούλιο να εκφραστεί επί των μέτρων. Ε, ρωτώ λοιπόν τι γίνεται με τους μηχανισμούς ελέγχου ε, και στο μέλλον εκτός από τις απλές διαμαρτυρίες που μπορούμε να εκφράσουμε μέσω των γνωμοδοτήσεών μας, τι άλλο μπορούμε να κάνουμε. Ευχαριστώ. Κάποιος άλλος θέλει το λόγο. Δεν θέλει κάποιο άλλο το λόγο, επομένω ε, η συγγήτρια, η κυρία Φλασίκοβα Μπένιοβα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κοιτάξτε, στην εισαγωγή που έκανα για την έκθεσή μου ανέφερα ότι η Επιτροπή οπωσδήποτε, η Επιτροπή μας εδώ οπωσδήποτε θα εκπονήσει γνωμοδότηση ακριβώς ε, για τα θέματα για τα οποία μέχρι τώρα ε, το Κοινοβούλιο δεν έχει δυνατότητα να μιλήσει. Ε, θα περιμένουμε τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων. Εάν εκεί δεν βρουν χώρο έκφρασης οι ανησυχίες μας, τότε θα τις αναφέρουμε αναφέρουμε σε δική μας γνωμοδότηση. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος, ευχαριστώ για την απάντησή σας. Δεύτερη ανταλλαγή απόψεων θα λάβει χώρα αργότερα. Αλλά ακόμα δεν έχουμε ορίσει προθεσμία υποβολής τροπολογιών. Κοιτάξτε, έχω την αίσθηση ότι θα πρέπει να διακόψουμε για λίγο, γιατί η κυρία Νατάσα Πίρκ Μουζάρ, η οποία είναι πρόεδρος του Κοινού Ποπτικού Οργάνου της Ευρωπόλ, δεν είναι εδώ. Ωραία λοιπόν. Να διακόψουμε μέχρι τις 9.30. 9.30 να ξαναείμαστε εδώ. Ευχαριστώ. Uh, Αγαπητοί συνάδελφοι, καλημέρα. Σήμερα θα ακούσουμε μια παρουσίαση της τρίτης έκθεσης επιθεώρησης κοινού υποπτικού οργάνου της Ευρωπόλ σχετικά με την υλοποίηση της συμφωνίας για το πρόγραμμα παρακολούθησης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Η παρουσία θα γίνει σήμερα από τη νέα πρόεδρο του κοινού υποπτικού οργάνου, την κυρία Πίρτς Μουσάρ, αν προφέρω σωστά το όνομά της. Κυρία Πίρτς Μουσάρ, θέλω να σα συγχαρώ και για την εκλογή σας και προσβλέπουμε στη μεταξύ μα συνεργασία. Νομίζω ότι θα σας δώσω όμως τώρα αμέσως το λόγο γιατί οι συνάδελφοι έχουν λάβει τα αρχικά συμπεράσματα, την έκθεση και περιμένουμε με ανυπομονησία να ακούσουμε την παρουσίασή σας. Κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ. Επιτρέψατε μου καταρχάς να σας ευχαριστήσω για τα καλά σας λόγια και τις ευχές σας πράγματι μόλις ε, ορίστηκα πρόεδρος του κοινού αποπτικού οργάνου της Ευρωπόλ ε, πριν από δύο εβδομάδες περίπου και είναι η πρώτη φορά που έχω την τιμή να σας παρουσιάσω το έργο του οργάνου αυτού. Και ελπίζω να στέφει με επιτυχία η προσπάθειά μας. Βέβαια, περιμένω και τις δικές σας ερωτήσεις. Ελπίζω να μπορέσω να δώσω απαντήσεις Στόχος του κοινού οργάνου της Ευρωπολ είναι ο έλεγχος του τρόπου με τον οποίο η Ευρωπόλ ε, χειρίζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τις βάσεις δεδομένων. Μία λοιπόν από τις αρμοδιότητες του κοινοποπτικού οργάνου είναι να επαληθεύσει κατά πόσον τα δεδομένα τα οποία διαβιβάζονται από την Ευρώπη στις Ηνωμένες Πολιτείες, διαβιβάζονται σύμφωνα με τους όρους της ε, συμφωνίας TFTP του προγράμματος παρακολούθησης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Θα σας παρουσιάσω την τρίτη έκθεση επιθεώρησης, δηλαδή είναι η τρίτη φορά που διενεργείται επιθεώρηση. Σε ό,τι αφορά την επιθεώρηση ενημερωθήκατε ως προς το τη συζήτηση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρώπης ε, εξακολουθεί, ε, είναι σε εξέλιξη και συζητείται και κατά πόσον η έκθεση αυτή η οποία είναι εμπιστευτική μπορεί να σας ε, παρουσιαστεί στα μέλη της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ καθώς και σε άλλα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θέλω να σας πω ότι στη χώρα μου τη Σλοβενία Είμαι υπεύθυνη και για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Επομένως, με την ιδιότητά μου αυτή γνωρίζω καλά την σχετική νομοθεσία. Την νομοθεσία δηλαδή που έχει να κάνει με την διαφάνεια των δεδομένων από τη χώρα μου αλλά και από άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δυστυχώς οφείλω να πω ότι δεν είμαι ικανοποιημένη. λόγω της εμπιστευτικότητας ε, της έκθεσης και ένα από τα καθήκοντα τα οποία ανέλαβα αφού το ανέλαβα τα καθήκοντά μου ως ε, πρόεδρος του ΚΕΟ είναι να πάρω αποφάσεις για το τι μπορεί να γίνει με αυτό το έγγραφο, την έκθεση επιθεώρησης. Δηλαδή μπορεί να δημοσιοποιηθεί ή όχι αυτό το έγγραφο. Αν λοιπόν έχετε ερωτήσεις σχετικά, με τα χαράς να σας απαντήσω. Να επανέλθω όμως ε, λίγο στην τρίτη αυτή έκθεση επιθεώρησης. Ένα από τα στοιχεία, μια πληροφορία που δίνεται, είναι ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε δεν μεταφέρουν έτσι, πολύ ακριβή δεδομένα μέσω του συστήματος SWIFT. Δεν είναι πολύ συγκεκριμένα τα στοιχεία. Και οι εξηγήσει που δίνουν σε ό,τι αφορά την επεξεργασία δεδομένων επίσης είναι ανεπαρκείς. Και αυτή είναι και μία από τις βασικές ε, επικρίσεις που ασκούμε. Η διαβίβαση δεδομένων συνεχίζεται. Πάντως, τα στοιχεία τα οποία συλλέγονται, διαβιβάζονται. Αυτό έχει διαπιστωθεί στη δεύτερη έκθεση επιθεώρησης και δεν δίνει νέα στοιχεία η τρίτη έκθεση επιθεώρησης πάνω σε αυτό. Μπορώ να σας πω όμως ότι οι ΙΠΑ δικαιολογούν καλύτερα τα αιτήματά τους και διαβιβάζουν περισσότερες πληροφορίες σήμερα. Οπότε, εν συνεχεία, η Ευρωπόλη έχει τη δυνατότητα να αξιολογήσει τις πληροφορίες αυτές. Πληροφορίες που είναι χρήσιμες για την Ευρωπόλη ώστε να δει ποια στοιχεία διαβιβάζονται και ποια όχι. Πρόοδος, λοιπόν, υπάρχει. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε ότι η αρχή της διαφάνειας δεν γίνεται σεβαστή, διότι το σύστημα SWIFT εξακολουθεί να διαβάζει όλα τα δεδομένα στο Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ. Και πρέπει να σας πω με κάθε ειλικρίνεια ότι ως νομικός αυτό το οποίο σημαίνει στην πραγματικότητα δυσκολεύομαι να το δεχθώ. Καθημερινά αντιμετωπίζω αυτά τα προβλήματα. Σας το λέω με κάθε ειλικρίνεια. Υπάρχει διάταξη, στην οποία υπάρχει και το σύστημα SWIFT, σύμφωνα με την οποία οι ΙΠΑ μπορούν να έχουν στη διάθεσή τους μόνο τα δεδομένα που είναι απολύτως απαραίτητα για να μπορέσουν να επιτελέσουν ε, το έργο του ελέγχου των δεδομένων. Και μέχρι εκεί. Καταλαβαίνετε τι θα πει αυτό από το πρίσμα της σύμβασης ε, τα ανθρώπινα δικαιώματα. Μόνο τα απολύτως απαραίτητα δεδομένα, όχι όλα τα δεδομένα. Άρα κανένας δεν μπορεί να με πείσει ότι είναι απολύτως απαραίτητο να διαβιβάζω όλα τα δεδομένα. Κάθε μήνα Ούτε ένα δευτερόλεπτο, αν θέλετε, δεν υπάρχει στη το του να μην πρέπει να διαβιβαστεί κάποιο δεδομένο. Καλύπτονται λοιπόν όλοι οι μήνες όλου του έτους από την υποχρέωση διαβίβασης δεδομένων, τα οποία δεδομένα στη συνέχεια αποθηκεύονται, φυλάσσονται για πέντε χρόνια στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η πρώτη λοιπόν διάταξη της συμφωνίας TFTP που πρέπει να γίνει γνωστή και στο Κοινοβούλιο, σε εσά ε, τους ε, βουλευτές, αλλά και ευρύτερα στην κοινή γνώμη. Είναι διάταξη η οποία προβλέπει μια προθεσμία τριών ετών προκειμένου να επαληθευθεί ποια ήταν η συμβολή των δεδομένων αυτών που διαβιβάστηκαν. Δηλαδή τι βοήθησαν να αποκαλυφθεί. Το θέμα είναι να υπάρχει αμοιβαιότητα. Τώρα, τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι αν η Ευρώπη διαβιβάζει δεδομένα προ τι ΗΠΑ αναμένει, όπω είναι φυσιολογικό, αντίστοιχα να διαβιβάζονται και από τη ΣΥΠΑ κάποια στοιχεία προ την Ευρώπη. Τι συμβαίνει όμω, Ξέρετε πόσε φορέ απέτησε η Ευρώπη από τι ΗΠΑ να διαβιβάσει κάποια δεδομένα. Μία και μόνο φορά, σα το απαντώ εγώ. Και τι θα πει αυτό. Θα πει ότι η Ευρώπη δεν είναι ικανή να καταπολεμήσει την τρομοκρατία ή μήπως σημαίνει ότι η Ευρώπη τελικά ζητά δεδομένα μόνο όταν αυτά είναι απολύτως απαραίτητα και αναγκαία ή μήπως σημαίνει ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε απαιτούν ζητούν υπερβολικά συχνά κάθε μέρα ε, στοιχεία, δεδομένα. Εσείς θα πρέπει να λύσετε το γρίφο αυτό. Εγώ δεν μπορώ να απαντήσω. Δεν μπορώ να σας δώσω τώρα μια τέτοια απάντηση. Και με αυτό θα ολοκληρώσω και την παρουσίασή μου. Είμαι, όπως είπα όμως, διατεθειμένη να απαντήσω στα ερωτήματά σας. Και εν είδη κατακλείδας να πω ότι στην τρίτη έκθεση επιθεώρησης λέμε ότι τελικά ε, προσκρούμε σε κάποιες πολιτικές αποφάσεις. Δηλαδή εμείς ως εμπειρογνώμονες, ως ειδικοί βρισκόμαστε σε ένα αδιέξοδο που λέγεται πολιτική. Εσείς οι Ευρωβουλευτές, εσείς οι Ευρωπαίοι πολιτικοί είστε αυτοί που θα πρέπει να λάβετε μια απόφαση ό,τι αφορά την έκθεση επιθεώρησης, η οποία θα πρέπει να δημοσιοποιηθεί τον Αύγουστο. Και θα πρέπει εσείς να κρίνετε κατά πόσο η συμφωνία TFTP πρέπει να παραμείνει αμετάβλητη ή αν πρέπει να τροποποιηθεί. Και αν το άρθρο 4 της λόγω συμφωνία ε, συμφωνίας πρέπει να αναθεωρηθεί. Μιλώ για το άρθρο που προβλέπει, βάσει το οποίο μάλλον προβλέπεται καθημερινή διαβίβαση δεδομένων από την Ευρώπη προς τις ΗΠΑ. Αυτά είχα να σας πω ως πρόεδρος του ε, κοινού εποπτικού οργάνου. Πρέπει να σας πω λοιπόν ότι μια πολιτική απόφαση είναι αυτή που τελικά θα πρέπει να ληφθεί. Αν θέλετε όμως την προσωπική μου άποψη, την άποψη μιας νομικού, αυτό δύσκολα μπορεί να γίνει αποδεκτό. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, σας ευχαριστώ θερμά. Διάβασα με μεγάλο ενδιαφέρον την έκθεση. Παρακολουθώ άλλωστε από την πρώτη ημέρα ε, το ζήτημα αυτό. Θα λάβω το λόγο, αφού όμως ε, προηγηθούν οι συνάδελφοί μου, να κάνω όμως μια παρατήρηση προκαταρκτικά. Βλέπω ε, την αίθουσα και ουσιαστικά απευθύνομαι σε αυτούς που λείπουν και σε αυτούς που είναι παρόντες. Πραγματικά, για τη συμφωνία SWIFT έγινε ολόκληρη ιστορία. Χρησιμοποιήσαμε για πρώτη φορά τις δυνάμεις που μας εκχωρήθηκαν από τη συνθήκη της Λισαβόνας και έχουμε ε, την ε, αρμοδιότητα ελέγχου. Πού είσαστε λοιπόν εσείς που δεν είστε εδώ, πού βρίσκονται όλοι. Έχουμε ε, αναλάβει την αρμοδιότητα κοινοβουλευτικού ελέγχου. Έπρεπε να πάρουμε πολύ σοβαρά το ρόλο μας πραγματικά. Από ό,τι υποδηλώνει τουλάχιστον η προσέλευση σήμερα. Για να δούμε ποιοι έχουν ζητήσει το λόγο. Σίπελ και μετά oh, So Σε λεπτό για να ε, βρει τα σλοβενικά η κυρία πρόεδρος του κοινοβουλευτικού οργάνου. Okay, go ahead. <laughs> Okay. Yeah, vielen Dank. Σας ευχαριστώ πολύ, πρόεδρε και ευχαριστώ και για τη σύντομη παρουσίαση της εκθέσεως. Πρέπει να πω ότι και εγώ αισθάνομαι δυσφορία για την συζήτηση που προηγήθηκε της αποφάσεως αυτής της συμφωνίας για το ενδιαφέρον της Επιτροπής μας στο θέμα αυτό. Όντως είναι πολύ μεγάλο, είναι κεντρική σημασία ζήτημα από την αρχή των εργασιών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν τηρήθηκαν οι αρχές που θα μπορούσαν να ικανοποιήσουν τις απαιτήσει μας και πέραν των όσων γράφονται στην έκθεση υπάρχουν και άλλα σημεία επίκρισης από πλευράς μας, τα οποία δεν λειτουργούν σωστά. Πιστεύω ότι είχαμε συνεννοηθεί ή ότι, αναζητήσαμε μία λύση από την αρχή για την συσταλτική θεώρηση για τον περιορισμό δηλαδή αυτών των δεδομένων που θα μεταφέρονταν, να μην είναι δυνατόν να περνάνε ανεξέλεγκτα τα προσωπικά δεδομένα. Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν φαίνεται να είναι διατεθειμένη να επεξεργαστεί κριτήρια με βάση τα οποία θα γίνεται η, η επεξεργασία των δεδομένων αυτών. Είναι πολλά δεδομένα τα οποία δεν προσφέρουν την ασφάλεια που θα θέλαμε στη μόρφη με την οποία μεταβιβάζονται και βλέπουμε ότι παρά το γεγονός ότι υπάρχουν και Ευρωπαίοι παρατηρητές στο US Treasury, ότι δεν υπάρχει δυνατότητα καλής συνεργασίας όπως θα θέλαμε. Και θα ήθελα να επισημάνω ότι με ενοχλεί ιδιαίτερο το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αφενός μας λέει όλα πάνε καλά, όλα βαίνουν καλώς, όλα λειτουργούν, αλλά παρόλα αυτά υπάρχουν κάποιες συστάσεις για να ε, προχωρήσουμε στην υλοποίηση και από την άλλη Εάν, ρωτάει, λέει η Επιτροπή ότι όλα αυτά λειτουργούν ε, κατά τρόπο απρόσκοπτο, γιατί μένουν εγκρυπτό και παραβίστο αυτά τα ε, στοιχεία και τα έγγραφα. Εγώ δεν λέω ότι θα πρέπει και οι 736 βουλευτές να πάρουν στα χέρια τους όλα αυτά τα έγγραφα, είναι απόρριτα και ότι θα πρέπει να διακινδυνεύσουμε την άλλη μέρα να βγουν στον τύπο. Αλλά δεν υπάρχει ε, δεν καταλαβαίνω γιατί δεν υπάρχει καμία δυνατότητα, καμία πρόσβαση, καμία ε, ενημέρωση. Γι' αυτό διερωτώ με τι είδου μυστικά κρύβουν αυτά τα έγγραφα που δεν μπορούμε ούτε εμείς εδώ μέσα στο κοινοβούλιο να έχουμε πρόσβαση. Και ω εκ τούτου περιορίζεται και η δυνατότητά μας στην πραγματικότητα, στην ουσία να εξετάσουμε αυτό το οποίο είναι και καθήκον μας, εάν δηλαδή η συμφωνία πληρεί τα συμπεφωνημένα, τα συμπεφωνηθέντα. Και ως εκ τούτου δεν μπορώ να είμαι αισιόδοξη, γιατί υπάρχουν κάποιες πληροφορίες που κυκλοφορούν για το πόσο καλά ή λιγότερα καλά μάλλον λειτουργεί όλο αυτό το σύστημα. Έχουμε υποβάλει ερωτήσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία απάντησε θα έλεγα κατά τρόπο χαρακτηριστικό. Ε, πάντως τα πράγματα δεν πάνε όπως τα περιμέναμε εδώ στο Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ κυρία Βέμπερ και μετά ο κύριος Ευχαριστώ πρόεδρε και ευχαριστώ πολύ κυρία Μουσάρ για την παρουσίαση σας. ψηφίζοντας υπέρ αυτής της συμφωνίας διδάχτηκα ένα πράγμα ότι δεν πρόκειται να ξαναψηφίσω ποτέ περιμένοντας να συμβούν θαύματα. Γιατί από ό,τι φαίνεται θαύματα δεν συμβαίνουν. Το αντίθετο μάλλον. Για τα πράγματα πήγαν δυστυχώς προς τα εκεί που φοβόμασταν ότι θα πάνε. Το μόνο καλό στοιχείο αυτής της συμφωνίας είναι το γεγονός ότι μπορέσαμε να δούμε ότι το μεικτό εποπτικό συμβούλιο της Europol ε, εργάζεται όπως όφιλε να εργάζεται και είχαμε τη χαρά να σας συναντήσουμε και να σας γνωρίσουμε. Αλλά πέραν αυτού, εγώ δεν λέω ότι θα πρέπει να ζητήσουμε περισσότερα ε, στοιχεία από τις ΗΠΑ, αλλά βλέπω ότι κάνουν ό,τι θέλουν. Βρήκανε τις πόρτες τις δικές μας ανοιχτές πολύ περισσότερο από ό,τι περιμένανε, ορθάνυχτες, και θα έλεγα ότι για τη δική τους την οπτική δεν είναι κατάχρηση αυτό που κάνουν. Το πρόβλημα που έχουμε εμείς έχει να κάνει με τις δικές μας αρχές. Γιατί όπως πολύ σωστά λέτε, εάν ο Ευρωπαίος μόνο άπαξ υποβάλλει το αίτημα, γιατί εμείς δεν καταπολεμούμε την τροποκρατία. Πρέπει να γίνεται όμως με τρόπο ε, σωστό το τι κάνουν όλα αυτά τα δεδομένα τα οποία αποθηκεύουν οι Αμερικανοί στους ηλεκτρονικούς τους υπολογιστές. Νομίζω ότι ξεπερνάει οτιδήποτε θα μπορούσε να φανταστεί η δική μας φαντασία. Και Έχω επίση ένα ερώτημα το οποίο θα μου πείτε είναι ρητορικό και το ξέρω, αλλά σε τελευταία ανάλυση πώ δουλεύουν τα πράγματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σα ακούσαμε τώρα με την ομιλία σα που μα είπατε ότι παρουσιάσατε, υποβάλατε μια έκθεση την οποία έχει επεξεργαστεί διεξοδικά το Εποπτικό Συμβούλιο, αλλά σε κάποιο άλλο σημείο εμφανίζεται ο κύριος Ράιτ για να πει κάτι τελείω διαφορετικό. Και περιμένω να ακούσω τι έχει να πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι κανεί εδώ από την Επιτροπή που να τολμά να πάρει το λόγο σήμερα και επιτροπή δεν εννοώ μόνο τον υπάλληλο της Επιτροπής, ανεξαρτήτως του ε, επίπεδου, ε, του, βαθμού που έχει, που θα είναι και πολύ ψηλό ίσως, αλλά εννοώ τον Επίτροπο, γιατί μιλάμε για πολιτική βούληση εδώ. Μπορώ να συνεχίσω έναν κατάλογο, γιατί έχουμε και δικούς μας ε, παρατηρητές στις Ηνωμένες Πολιτείες για να εποπτεύουν, να παρακολουθούν. Πότε είδαμε κάτι το ουσιώδες από τους δικούς μας, τους υπαλλήλους που τελευταία ανάλυση πληρώνει ο Ευρωπαίος ε, φορολογούμενος. Γιατί δεν μπορούμε κάποια στιγμή να κάτσουμε όλοι μαζί και να τα συζητήσουμε. Δεν χρειάζεται να απευθύνουμε κατηγορίες ή να προβάλλουμε ε, δικαιολογίες και άμυνα. Αλλά έχουμε να κάνουμε ένα θέμα πάρα πολύ σημαντικό για τους πάντες. Και θα έλεγα ότι είναι Στη τελευταία ανάλυση περί τι διασπάθηση χρημάτων το να κάνουμε συζήτηση χωριστά με τον κάθε φορέα κάθε φορά. Και έχω μια ερώτηση, η οποία δεν θα ήθελα να φανεί αγενής, αλλά παρακαλώ, θα ήθελα να μάθω. Με την Επιτροπή, με την Επιτροπή, με την Επίτροπο Μάλστρομ, συζητήσατε τα πορίσματα αυτά. Και αν ναι, Πώ αντέδρασε στη συζήτηση αυτή η κυρία Μάλστρομ. Ελπίζω ότι και εμεί θα έχουμε την ευκαιρία να τη δούμε. Όπω είπαμε, όχι σήμερα, ε, ο καθένα με τη σειρά του, εν πάση περιπτώσει, αλλά... Και ξέρω ότι είστε πολύ νέα στη θέση αυτή, αλλά από προηγούμενε συνομιλίε του, Συμβουλίου με την, ε, του Εποπτικού Συμβουλίου με την Επίτροπο Μάλστρομ. Τι έχετε να μα πείτε. Ευχαριστώ κύριε thank... Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Μουσάρα για την εξαίρετη έκθεση που μας έκανε, μεταφέροντάς μας ε, τι, όλα αυτά που συμβαίνουν, τα οποία φυσικά δεν με ικανοποιούν. Δεν θα επαναλάβω αυτά τα οποία είπαν ήδη οι προραλήσασες ε, συνάδελφοι. Θα πω απλά ότι η δική μου πολιτική ομάδα, βασιζόμενη και σε αυτά που ακούσαμε σήμερα, αλλά και στα όσα υποπτευόμαστε από πριν, θα εργαστεί έτσι ώστε να σταματήσει ε, ε, το πρόγραμμα αυτό, κυρίως ε, τουλάχιστον όσον αφορά και το άρθρο 4 και σε σχέση και με αυτά που θα πρέπει να απαντήσει η κυρία Μουσάρα για την ερώτηση της κυρίας Βέμπερ, δηλαδή κατά πόσον έχει συζητήσει τα ευρήματα αυτά, τα πορίσματα με την Κομισιόν και ποια είναι η άποψη, η θέση της Κομισιόν. Αλλά εν κατακλείδη εμείς δεν είμαστε ικανοποιημένοι και επομένως ε, θα προσπαθήσουμε να σταματήσουμε την αναθεώρηση του άρθρου 4. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Μπάουερ. Αυτή η κατάσταση είναι λίγο περίεργη, περίπλοκη. Ε, αναφέρομαι στη δική μας κατάσταση γιατί συζητούμε για μια γνωμοδότηση την οποία δεν έχει ακόμα διαβάσει κανένας. Και Έχουμε κάποιες ε, πληροφορίες ε, οι οποίες όμως ακόμα δεν έχουν διακριβωθεί, δεν έχουν επαληθευτεί. Ακούσαμε από την κυρία Μουσάρ ότι, πρόκειται για, ότι υπάρχουν αρχές οι οποίες δεν έχουν γίνει σεβαστές ε, τα, κράτη, ε, τα, τα, οι Ηνωμένες Πολιτείες ε, κρατούν όλα τα στοιχεία επίσης δεν έχουν γίνει σεβαστές οι αρχές της, του απορρίτου και της εμπιστευτικότητας αναρωτιόμαστε όμως υπάρχει δυνατότητα να αλλάξει ας πούμε η σύμβαση νομικά πιστεύουμε ότι δεν, ε, ε, η σύμβαση αυτή δεν είναι σωστή, άρα μπορεί να τροποποιηθεί. Ευχαριστώ πολύ. Κάποιος άλλος, όχι. Ε, πρώτον, νομίζω να... Θα απαντήσω εγώ μάλλον δύο ερωτήσεις που απευθύνατε, κυρία Μπάουερ. Ε, το έγγραφο είναι δημόσιο και η γραμματεία το έχει κυκλοφορήσει, είναι διαθέσιμο, είναι πολύ σύντομο, δύο-τριών σελίδων. Δεύτερον, το θέμα της ε, συνθήκης, ε, περί αυτού πρόκειται και γι' αυτό έγινε όλη η συζήτηση. Τώρα μπορούμε να ζητήσουμε από την Κομισιόν ε, να προχωρήσει σε πρόταση για την ανέρεση της συμφωνίας, αλλά δεν μας ακούει, κοφεύει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στην ουσία δηλαδή, ε, εντάξει μπορούμε να ζητήσουμε για ενέργεια της ε, συμφωνίας, αλλά δεν είναι πλέον η μπάλα στα δικά μας χέρια. Το, την πετάξαμε την μπάλα στο ε, γήπεδο της Κομισιόν. Κοιτάξτε, αυτό άλλωστε είναι ένα ζήτημα το οποίο το έχω παρακολουθήσει πάρα πολύ στενά. Ε, όπως ξέρουν και συνάδελφοι, έχω αναμειχθεί και με κάποιες διαδικασίες οι οποίες ζητούν πρόσβαση σε κάποια άλλα έγγραφα, κυρίως ε, το, την περσινή έκθεση που ξέρουμε ότι έχει ε, δημοσιευθεί. Ίσως πρέπει να δούμε ποιες είναι και οι διαδικασίες ε, για την ιεράρχηση των εγγράφων. Ε, για τη διαβάθμιση των ε, εγγράφων. Ε, νομίζω ότι για οποιαδήποτε αλλαγή πρέπει να πάμε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και αν φτάσουμε ενώπιον του δικαστηρίου μπορεί να περιμένουμε χρόνια μέχρι να βγει απόφαση αλλά αυτό δεν είναι καθόλου υπέρ της διαφάνειας. Επίσης πρέπει να πω ότι η στάση της Κομισιόν στο θέμα που μας απασχολεί δεν είναι σωστή. Αντί να ξεκινήσουν μία σε βάθος συζήτηση, στην ουσία ε, ε, κατηγόρησαν ε, ένα μέλος της ομάδας ότι είχε σύγκρουση συμφερόντων, που πιστεύω ότι ήταν μία απαράδεκτη στάση και μία απαράδεκτη κατηγορία και δεν πρόθεσε καθόλου την συζήτηση. Ελπίζω ότι αυτό θα διευθετηθεί. Βεβαίω, το κυριότερο σημείο εδώ, το πυρηνικό σημείο, ο κύριος στόχος, αν όχι ο μόνος στόχος της Συμφωνία SWIFT, είναι ε, να σταματήσει αυτή η χίδιν ε, μεταφορά δεδομένων. Και στην ουσία εσείς επιβεβαιώσατε αυτά που υποψιαζόμαστε, δηλαδή ότι ε, αυτό είναι αδύνατο να γίνει λόγω της φύσης του εγχειρήματο. Στην ουσία είπατε ότι αν αυτό ισχύει, αν αυτό είναι αληθές, τότε οπωσδήποτε θα έπρεπε να αναιρεθεί ή και να καταργηθεί η συμφωνία και επομένως εν τέλει να ακούσουμε από την Κομισιόν. Ένας από τους λόγους που και εγώ και άλλοι ψηφίσαμε για την, την ε, συμφωνία με μεγάλο δισταγμό είναι γιατί υποσχέθηκε η Κομισιόν ε, να αρχίσει να ε, συζητάει για την εξέβρεση ενός συστήματος ανάκτησης επιλεκτικής δεδομένων και όχι χίδιν μεταφοράς δεδομένων. Κοιτάξτε, πρόκειται για ένα απλό λογισμικό. Εάν το έχουν οι Αμερικανοί, γιατί δεν το έχουμε κι εμείς, γιατί ακόμα περιμένουμε, γιατί δεν μπορούμε να το έχουμε κι εμείς και κάτι άλλο. Αλλά βεβαίως αυτό αφορά απόφαση που πρέπει να, αποφασίσει να λάβει η Επιτροπή μας εδώ. Νομίζω, νομίζω ότι πλέον είναι επίγον να έχουμε απαντήσεις από πολιτικούς υπευθύνους. Πρέπει να έρθει κάποιος επίτροπος εδώ ή επίτροπος μάλλον να έρθει εδώ. Ζητήσαμε και μα είπε η Κομισιόν ότι ο κύριος Μανσαβίση μπορεί να έρθει ε, και να μας μιλήσει. Όχι, δεν μας αρέσει. Δεν μας αρέσει, δεν μας ικανοποιεί, δεν είναι αρκετό. Κοιτάξτε, έχει γίνει πολλή συζήτηση και αν δείτε ε, τι λόμπινγκ έλαβε χώρα έτσι ώστε να πιστεί η Κομισιόν, καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το ζήτημα. Ε, κατηγορηθήκαμε μάλιστα ότι δημιουργήσαμε ένα κενό ασφαλείας, security gap, Τώρα είναι σαφές πλέον ότι η συμφωνία ε, θα μπορεί να εφαρμόζεται πλέον ε, καλύτερα από ό,τι στην αρχή. Αλλά πέραν της καλής ή κακής ε, υλοποίησης, η ίδια η συμφωνία είναι κακή. Και δεν έχουν επιτευχθεί οι στόχοι της Διατλαντικής Συμφωνίας. Το ζήτημα της διαφάνειας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι το μεγαλύτερο νομίζω. Όλη αυτή η διαδικασία ε, της διαβάθμισης ε, είναι μάλλον ερμητική, δεν είναι καθόλου καθαρή. Μεταφέρονται μαζικά στοιχεία στην, ε, στις ΗΠΑ και μπορεί αργότερα να κάνουμε συμφωνία και με μια άλλη χώρα και τότε να, δίνουμε όχι μόνο τα στοιχεία των ταξιδιωτών αλλά ας πούμε και τα στοιχεία των τον και τα τραπεζικά μας στοιχεία των πολιτών μας. Υλοποιείται λοιπόν μια συμφωνία ε, και τελικά δεν έχουμε καμία πρόσβαση σε όλη αυτή τη διαδικασία. Ε, ε, στην ουσία εμείς εδώ προσπαθούμε να υπεραμεινθούμε των δικαιωμάτων των πολιτών γιατί στο τέλος τέλος αυτονών των πολιτών τα στοιχεία μεταβιβάζονται. Εν πάση περιπτώσει, εμεί σα ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε εδώ και κάνετε την παρουσίαση αυτή. Θα δώσω το λόγο στην Κομισιόν και ελπίζω ότι θα πάρουμε κάποιε ικανοποιητικέ απαντήσει. Επαναλαμβάνω πάντω ότι η Επιτροπή μα και φαντάζομαι ελπίζω να συμφωνείτε μαζί, μας, μαζί μου, ε, θα πρέπει οπωσδήποτε επιγόντω να καλέσει την κυρία Μάλστρομ, την Επίτροπο Μάλστρομ, όχι τον κύριο Μασαβίζη ή κάποιον άλλον υψηλό βαθμό αξιωματούχο, την κυρία ε, ε, Επίτροπο έτσι ώστε να μπορέσει να λυθεί το ε, πρόβλημα. Θα καλέσω την ε, Κομισιόν να απαντήσει και σε κάποια ερωτήματα και μετά να σας δώσω τον λόγο κυρία Μουζάρ για, την, ε, για το τέλος της παρουσίασής σας. Ο κύριος Λόξ και η κυρία Μαγιόν. κύριος Λόξ. Καλημέρα σας. Θα προσπαθήσω να απαντήσω, αν και είμαι ένας ταπεινός ε, υπάλληλος. Νομίζω ότι είναι δύο αυτά τα οποία συζητούμε κυρίως εδώ. Το πρώτο, η τρίτη έκθεση επιθόρησης του κοινοποπτικού οργάνου που δημοσιεύθηκε πριν από κάποιους μήνες. Εγώ νόμιζα ότι περί αυτού θα συζητούσαμε σήμερα. Ποια είναι τα πορίσματα και ποιες είναι οι συστάσεις αυτής της έκθεσης. Υπήρξαν όμως ευρύτερα ζητήματα για την καταλληλότητα, την αποτελεσματικότητα και την όλη λειτουργία της συμφωνίας ε, TFTP. Τα τέθηκαν. Ας συζητήσουμε όμως πρώτα το ζήτημα το πρώτο, δηλαδή την ε, τρίτη έκθεση επιθεώρησης του κοινού εποπτικού οργάνου. Και θα δώσω κάποιες απαντήσεις. Η τρίτη έκθεση επιθεώρησης σημειώνει και καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η Ευρωπόλ ουσιαστικά πλέον εκτελεί τα καθήκοντά της με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και αυτό κυρίως χάρη ε, στους ανθρώπους της προστασίας δεδομένων που εξετάζουν πάρα πολύ προσεκτικά όλα τα σχετικά θέματα. Αυτό το λέει η τρίτη έκθεση μας, μας ικανοποιεί αυτό. Μας ικανοποιεί επίσης και θα ε, συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με τους συναδέλφους μας από το κοινό εποπτικό όργανο, διότι πιστεύουμε ότι αποτελούν μια σημαντική προστιθέμενη αξία για την όλη διαδικασία. Αυτό είναι μια ε, σταθερή πεποίθηση της ε, Επιτροπής ότι είναι σημαντική η προστασία των δεδομένων και θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με το ΚΕΟ. Να πω επίσης ότι ο κύριος Μανσεβίζη πράγματι όταν ε, μάλλον ε, συναντήθηκε με τον επικεφαλή της Επιτροπής για το άρθρο 21 και με κάποιους άλλους αρμοδίους και νομίζω ότι πλέον ε, είναι σαφή τα πράγματα. Θέλουμε νομίζω να έχουμε μια καλή συνεργασία και έχουν τεθεί βάση προς αυτό. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη διαβάθμιση, πρέπει να σας πω ότι η διαβάθμιση γίνεται από το συντάκτη ενός εγγράφου και κανέναν άλλον. Ο μόνος ε, άνθρωπος ή φορέας που αποφασίζει ε, για το αν ένα έγγραφο είναι ε, διαβαθμισμένο σε ποια, και σε ποια κατηγορία, ο μόνος που αποφασίζει είναι ο συντάκτης. Το ΚΕΟ αποφάσισε στην προκειμένη περίπτωση τη διαβάθμιση, όχι η Ευρωπόλ, όχι η Κομισιόν. Και αυτό πρέπει να το έχετε υπόψη για να καταλάβετε. Από τη στιγμή που διαβαθμίζεται ένα έγγραφο, φυσικά υπάρχουν κανόνες για την ε, από ε, διαβάθμιση, για την ε, δημοσιοποίηση δηλαδή. Και πάλι την τελική απόφαση τη λαμβάνει συντάκτη του εγγράφου. Υπάρχουν όμω ε, κάποιε παράμετροι νομικέ και διαδικαστικέ που πρέπει να ληφθούν υπόψη και σε ανταλλαγή επιστολών τα συζητήσαμε αυτά. Για να μπορεί λοιπόν να δημοσιοποιηθεί ένα έγγραφο πρέπει να αντιμετωπιστούν κάποια εμπόδια τότε δεν υπάρχει ικανοποιητική ε, και εύρυθμος λειτουργούσα ε, ρύθμιση, ε, αυτό δημιούργησε τα προβλήματα. Εγώ δεν είμαι υπεύθυνο και ούτε θα δώσω διαφθουσμένες πληροφορίες σε ανθρώπους που δεν έχουν άδειες, που δεν έχουν εγκρίσεις ασφαλείας και που δεν έχουν ουσιαστικά δικαίωμα πρόσβασης. Από εκεί και πέρα, εξίσου σημαντικό είναι το θέμα ότι στην κοινότητα ε, intelligence, ανταλλαγής πληροφοριών, ε, υπάρχουν κανόνες. Θα πρέπει να δοθεί συγκατάθεση, συνένεση ενός τρίτου, σε περίπτωση που οι πληροφορίες ανήκουν σε έναν τρίτο, προτού δημοσιοποιηθούν οι πληροφορίες. Θα πρέπει δηλαδή για την αποκάλυψη, τη δημοσιοποίηση των πληροφοριών να συνενέσει ε, το τρίτο μέρος. Οι αρχές των ΗΠΑ αποφάσισαν στην προκειμένη περίπτωση να μην το πράξουν λόγω του επιχειρησιακού χαρακτήρου ορισμένων στοιχείων. Πρόεδρος, να σας διακόψω, διότι δεν μιλάμε για τη διαφάνεια. Υπάρχει και ο εξή κανόνας. Θα πρέπει κάθε διαβάθμιση να αιτιολογείται συγκεκριμένα και λεπτομεριακά. Το να διαβαθμίσετε ένα ολόκληρο έγγραφο που λέτε ότι έχει επιχειρησιακές πληροφορίες, το να το διαβαθμίζουμε όλο το έγγραφο αυτό δεν μπορεί να είναι αλήθεια ο εκπρόσωπο τη Κομισιόν. Μα δεν το αποφασίσαμε εμεί. Δική του επιθεώρηση ήταν δική του έκθεση. Το κοινό υποπτικό όργανο αποφάσισε να είναι ε, εμπιστευτικό το έγγραφο αυτό. Είναι δική του έκθεση. Δεν το κάναμε εμεί. Δεν το αποφασίσαμε εμεί αυτό. Τώρα έρχομαι στα ευρύτερα ζητήματα και ερωτήσεις. Να πω καταρχά ότι σέβομαι απόλυτα τι απόψει σα και τις ερωτήσεις και αμφιβολίες που έχετε για τη συμφωνία TFTP. Δεν ήρθα εδώ για να επεκταθώ πάνω σε αυτό. Αυτό που θέλω να πω είναι το εξής. Η τελευταία ε, συνολική ε, εκτίμηση της ε, αποτελεσματικότητας και καταλληλότητας του προγράμματος και της συμφωνίας TFTP έχει εκδοθεί τον Δεκέμβριο στη δεύτερη έκδοση της Γενικής Αξιολόγησης από την Κομισιόν, από την αρμόδια αρχή, τον είπα και από τη, τον αντιπρόεδρο της Eurojust και από την ε, Ολλανδία και το Βέλγιο, από εκπροσώπους. Μια κοινή αξιολόγηση έγινε δηλαδή και καθίσαμε να συζητήσουμε όλοι και με το Υπουργείο Οικονομικών, ε, με την Ευρωπόλ, ε. Έγινε λοιπόν μια κοινή επιθεώρηση και σε αυτή την έκθεση περιλαμβάνεται η εκτίμηση ότι αφού τέθηκε σε ισχύ η συμφωνία και σταδιακά έχουμε αυτά τα χέρια και τι ασφαλιστικέ δικλίδες, πλέον λειτουργεί ικανοποιητικά η συμφωνία, πολύ ικανοποιητικά. Παναλαμβάνω όμως ότι ούτε εγώ ούτε η Κομισιόν μόνο κάναμε αυτή την εκτίμηση. Είναι ένας μεικτό φορέας αυτός που προέβησε αυτή την εκτίμηση. Φυσικά και επαγρυπνούμε Φυσικά και επιβλέπουμε την κατάσταση. Είμαστε σε συνεχή επαφή με τις Αμερικανικές Αρχές και την Ευρωπολ ώστε πραγματικά να ισχύουν και να εφαρμόζονται αυστηρά οι ασφαλιστικές δικλίδες. Θέλω να σας πω ότι το άρθρο 6, πράγματι, το άρθρο 6 της Συμφωνίας TFTP προβλέπει ότι μετά από τρία χρόνια από την ε, έναρξη ισχύω η Κομισιόν θα αναθεωρήσει ή θα επανεξετάσει την συμφωνία ε, στο σύνολό τη. Και πράγματι θα το πράξουμε φέτο το καλοκαίρι. Σύστημα εξαγωγή δεδομένων υπάρχει, λέει πρόεδρο. Ναι, πράγματι, όπω γνωρίζετε, τον Ιούλιο του 2011, ένα χρόνο φτέθηκε σε ισχύ συμφωνία. Αυτό το πρώτο έτος εφαρμογής ε, το χρησιμοποίησαμε ως έτος αναφοράς και επίσης κάναμε αναλύσεις, ε, είχαμε και διαβουλεύσεις με πολλούς ε, ενδιαφερομένους φορείς και έχουμε δημοσιοποιήσει το λεγόμενο option paper, μια ανακοίνωση δηλαδή της ε, Κομισιόν που παρουσιάζει τις επιλογές για ένα σύστημα ευρωπαϊκό. Έγιναν συζητήσεις και στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο με τις Final Investigation Units με όλους τους εμπλεκομένους φορείς και ολοκληρώνουμε την μελέτη επιπτώσεων για να δούμε τα υπέρ κατά ε, τις ε, διάφορες ε, διατυπώσεις και ό,τι άλλο χρειάζεται. Η πρώτη έκθεση μελέτης επιπτώσεων έχει καταρτιστεί αλλά μας ζητήθηκε να το επεξεργαστούμε το κείμενο αυτό και σε αυτή τη φάση βρισκόμαστε. Θέλουμε να το χτενίσουμε, αν θέλετε, ε, το κείμενο της ε, μελέτης αυτής επιπτώσεων. Και βέβαια θα διαβιβάσω την πρόσκλησή σας στην κυρία Μάλνστρομ. Πρόεδρε, κύριε Λόξ, σας σέβομαι και γνωρίζω επίσης ότι δεν εκφράσετε προσωπικέ σα απόψει αλλά απόψει τη Κομισιόν. Να σα πω όμω ότι δεν απαντήσατε στο ερώτημα. Ουσιαστικά πράγματι υπήρξε η δημοσιοποίηση αυτή τη ανακοίνωση από την Κομισιόν, αλλά αυτό δεν αφορούσε την εξαγωγή δεδομένων πρωτού σταλούν στη ΣΥΠΑ, αλλά αφορούσε την αποθήκευση δεδομένων στην Ευρώπη. Αυτό είναι ένα εντελώς διαφορετικό σύστημα. Εγώ σα μιλάω για ένα απλό λογισμικό. Αυτό που χρησιμοποιούν οι Αμερικανοί για να φιλτράρουν τα δεδομένα. Θα μπορούσαμε να έχουμε το ίδιο λογισμικό. Τρία χρόνια μετά δεν έχω απάντηση γιατί δεν το έχουμε αυτό το λογισμικό. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα σχόλιά σας για τη δεύτερη κοινή αξιολόγηση που είπατε πόσο ικανοποιημένοι ήταν όλοι, τι να σα πω, εγώ νομίζω ότι θυμάμαι ότι τα μέλη αυτής της κοινή ομάδας δεν είχαν πρόσβαση πρώτα απ' όλα σε όλε τι πληροφορίε. Και δεύτερον, δεν ήταν τόσο ικανοποιημένα όλα τα μέλη. Υπήρξαν αφισβητήσεις, υπήρξαν ενστάσεις Αυτέ είναι παρατηρήσεις παρατηρήσει μου. Ε, στις συζητήσεις αυτές τελικά βλέπω να επαναλαμβάνουμε τα ίδια και τα ίδια και να μην έχουμε απαντήσεις από την Κομισιόν. Θα στραφώ όμως τώρα στην κυρία Μουσάρ για να μας δώσει τις δικές της καταληκτικές παρατηρήσεις. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρίες και κύριοι βουλευτές. Σας ευχαριστώ για τις ερωτήσεις σας. Ευχαριστώ και τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα πάρω τις ερωτήσεις με τη σειρά. Καταρχάς, για τη δήλωση του εκπρόσωπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μας πετάξατε το μπαλάκι. Είπατε ότι εμείς κάνουμε τη διαβάθμιση ως απορρίτων των εγγράφων. Πρέπει να πω με απόλυτη ειλικρίνεια ότι ε, ως ε, πρόεδρος εδώ και μισή μήνα αυτού του μεικτού εποπτικού συμβουλίου. Πάντοτε υποστηρίζω, υποστήριξα ότι δεν έπρεπε να είναι απόρριτη αυτή η έκθεση, τουλάχιστον όχι στο σύνολό της. Έχω ένα χρόνο τώρα ε, απασχόληση στον χώρο αυτόν και έχουμε εκπροσώπους των κρατών μελών, στα οποία κράτη-μέλη βεβαίως ισχύουν και διαφορετικοί νόμοι. Εμείς στη Σλοβενία έχουμε μια πολύ καλή νομοθεσία για την δυνατότητα πρόσβασης ε, σε απόρριτα έγγραφα από το κοινό. Εγώ λοιπόν έχω μια πολύ πιο θετική στάση απέναντι στη διαφάνεια και θεωρώ ότι θα πρέπει τα έγγραφα να είναι δημόσια χωρίς καν να χρειάζεται να υποβληθεί αίτηση. Ε, ως εκ τούτου λοιπόν καθήκον μου, στη θέση αυτή που ανέλαβα, θεώρησα να συνεχίσω και γι' αυτό ρώτησα και στην ε, Europol εάν το έγγραφο αυτό μπορεί να διαβαθμιστεί ως μη απόρριτο. Πάντοτε διαβαθμιζόταν ως ε, απόρριτο γιατί ε, περιελάμβανε στοιχεία, δεδομένα, τα οποία ε, ήταν απόρριτα, τα στοιχεία δηλαδή που είχαν συλλεγεί κατά τις ε, επιθεωρήσεις και γιατί σεβαστήκαμε και το γεγονός ότι τα κράτη-μέλη μπορεί να πούν ότι δώσαμε απόρριτα στοιχεία και ως εκ τούτου αν αυτά συμπεριληφθούν σε ένα έγγραφο θέλουμε και το έγγραφο που θα περιλαμβάνει τα δικά μας στοιχεία τα εθνικά να είναι απόρριτο. Αυτό σεβόμαστε. Αλλά από την άλλη η θέση μας, η πάγια θέση μας είναι και η κυρία Ινετφέλτ το είπε η θέση μας λοιπόν είναι ότι ποτέ δεν πρέπει να επιμένουμε να επιβληθεί απόρριτος χαρακτήρας στο σύνολο του εγγράφου. Εφόσον περιλαμβάνονται δημόσια γνωστές πληροφορίες, τότε έστω μερική πρόσβαση, partial access, πρέπει να υπάρχει στο έγγραφο. Και πρέπει να πω ότι διάβασα το έγγραφο διεξοδικά, δεν υπάρχει τίποτα το απόρριτο μέσα. Εάν ήταν στο δικό μου χέρι δηλαδή θα είχα εδώ και πολύ καιρό ε, δημοσιεύσει, κοινοποιήσει το έγγραφο αυτό. Εδώ βρισκόμαστε σε ένα φαύλο κύκλο ουσιαστικά. Γίνονται τα αιτήματα στην Europol, η Europol επιληθεύει αν θα πρέπει να δημοσιευθούν τα έγγραφα, ε, πρέπει να ρωτήσουμε τον ε, τρίτο εταίρο, εν προκειμένου Ηνωμένες Πολιτείες, εάν έχει καμία αντίρρηση και αν θα πρέπει να παραμείνει σε διαβάθμιση απορρίτου το έγγραφο. Ενάμιση χρόνο τώρα γυρνάμε γύρω-γύρω και δεν κάνουμε τίποτα. Λένε όχι οι Αμερικανοί, λέει αναγκαστικά όχι η Europol και το καθεξής. Καθήκον μου λοιπόν εγώ θεώρησα από την ανάληψη των ε, αρμοδιότητων αυτών και σας διαβεβαιώ ότι θα το κάνω μέχρι κάθε ε, τελευταία δυνατότητα να επαληθεύω την δυνατότητα δημοσιοποίησης του εγγράφου. Να μην είναι δηλαδή βαθμισμένο ως απόρριτο 100%. Όσο υπάρχει αυτό θα το επαληθεύω εγώ αν υπάρχει κάποια δυνατότητα, κάποια διαδικασία η οποία θα μου επέτρεπε να το διαβαθμίσω ως μία απόρριτο θα το έκανα. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει και να τηρήσουμε τις γενικές διατυπώσεις, δηλαδή να ρωτήσουμε τον τρίτο, την τρίτη πλευρά, τη λεγόμενη του Αμερικανούς, οι οποίοι όμως λένε, εν προκειμένου, όχι. Μη αιτιολογημένη απάντηση πρέπει να πω, νομικά δηλαδή δεν είναι αιτιολογημένη η αρνητική απάντηση. και άρα θα πρέπει να ξέρω επακριβώς ποια είναι τα απόρριτα εκείνα στοιχεία τα οποία εντοπίζονται και τα οποία θα πρέπει να καταστήσουν απόρριτο το έγγραφο στο σύνολό του. Εγώ νομίζω ότι πλέον θα πρέπει να αναλάβουμε την ευθύνη στα δικά μας χέρια και να λάβουμε μόνοι μας την απόφαση. Ιδάλλως, όπως είπε ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είναι απόρριτο και παραμένει Απόρριτο. Αλλά αυτό θα είναι το δικό μου καθήκον να αμφισβητήσω αυτές τις επιλογές. Ο κύριος από την Επιτροπή είπε ότι στην πράξη λειτουργεί πολύ καλά αυτή η συμφωνία. Ναι, λειτουργεί πολύ καλά, δίνουμε ό,τι μας ζητάνε αλλά ίσω θα πρέπει να κάνω μία εξήγηση τώρα για το πώ δίδονται τα στοιχεία αυτά. Κάνει το αίτημα η αμερικανική πλευρά ε, μέσω του SWIFT. Πρέπει να επαληθεύσει όμω τη συμφωνία Europol από τη, για να ε, βεβαιωθεί ότι είναι στοιχεία αυτά τα οποία μπορούν να διατεθούν στην αμερικανική πλευρά. Τουλάχιστον αυτό θεωρώ ότι είναι το δικό μα καθήκον. Τότε τα πάντα τα στοιχεία στην, στο SWIFT και από το SWIFT στους Αμερικανούς. Εμείς λοιπόν από πλευρά μας ως Εποπτικό Συμβούλιο, πέραν αυτού δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο. Παρά μόνο αυτά που ορίζει το σημείο 6 της, ή το άρθρο 6 της συμφωνίας. Νομίζω ότι θα πρέπει όμως και να είναι κανείς πιο θαραλέος και να αμφισβητήσει αυτές τις επιλογές. Γιατί να είναι η Europol κομμάτι αυτού του συστήματος, γιατί είναι ο τρίτος πυλώνας συστήματο η Europol. Μόνο το γραμματοφορέα θα, θα παριστάνει τον ταχυδρόμο. Δεν θα πρέπει να επαληθεύει σωστά, με ακρίβεια, εάν τα στοιχεία που συντρέχουν, που απαιτείται, όντως συντρέχουν. Εγώ θεωρώ ότι αυτή πρέπει να είναι η δουλειά της Europol και πρέπει να την επιτελεί ε, με θάρρος, με παρησία. Γιατί αυτός ο οποίος έχει και το δικαίωμα, να έχει μάλλον το καθήκον να αποστέλει τα στοιχεία, πρέπει να έχει και το θάρρος να πει όχι δεν τα αποστέλνω. Διότι δεν είναι σύμφωνα με, την, ε, με τις ε, διατάξεις ή διαφορετικά. Είμαστε η αδύναμη πλευρά, ο αδύναμος εταίρος της συμφωνίας. Οπότε θα πρέπει να το ξανακοιτάξουμε. Δεν νομίζω ότι το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι όμω να γράφουμε καταβατικά σε οποιοδήποτε αίτημα τη άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Βεβαίω και αντιλαμβάνομαι πόσο σοβαρό είναι ο αγώνα για την ε, καταπολέμηση τη τρομοκρατία. Βεβαίω και αντιλαμβάνομαι ότι θα πρέπει να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μα. Αλλά και στην πατρίδα μου τη Σλοφενία, έχουμε τέτοια ζητήματα. Η αστυνομία, οι μυστικές υπηρεσίες είναι υποχρεωμένες να εκτίθενται, να ε, συλλέγουν στοιχεία κτλ. Αλλά δεν είμαστε υποχρεωμένοι να εκτιθέμεθα σε ε, εσφαλμένες επιλογές. Εν πάση περιπτώσει, εγώ δεν μπορώ να μιλήσω περισσότερο για θέματα πολιτικά, γιατί ο τομέας μου είναι νομικός είμαι, είναι άλλο ο τομέας μου, αλλά όπως είπα, ίσως θα πρέπει κάποια στιγμή να ληφθεί μία απόφαση για το αν θα γίνεται δημόσια γνωστό το έγγραφο. Εγώ ως υπεύθυνη για ενημέρωση ξέρω πολύ καλά ε, τι σημαίνει διαβάθμιση ως απορία του ενός εγγράφου. Ξέρω ότι υπάρχει δυνατότητα της μερικής διαβάθμισης. Συμβαίνει και στη Σλοβενία αυτό, το έχουμε υπόψη μας. Επομένω, νομίζω ότι είναι δυνατόν να γίνει. Καταρχά, και τώρα να περάσω στι ερωτήσει των συναδέλφων, των βουλευτών. Κυρία Μπάουερ, καταρχά. Με ρώτησε η κυρία Μπάουερ, λοιπόν, εάν ε, ξέρω, γνωρίζω και άλλε περιπτώσει μη σεβασμού τη αρχή τη ε, αμοιβαιότητα. Δεν μπορώ να πω τίποτα, γιατί ε, η μεταβίβαση δεδομένων οποιαδήποτε στιγμή αποτελεί πρόδειλο αποτέλεσμα και αυτό ε, εμένα που είμαι νομικός μου δημιουργεί πρόβλημα. Με ρωτάτε αν πρέπει να αλλάξει κάτι. Ως πρόεδρος του κοινού υποπτικού οργάνου θα επιθυμούσα να τροποποιηθεί ε, η ε, συμφωνία, κυρίως το άρθρο, ε, το οποίο αφορά την τροποποίηση διαχείρισης δεδομένων. Αυτή η συμφωνία σήμερα δεν μας δίνει σαφείς ενδείξεις πότε μπορούμε να απαντήσουμε θετικά και πότε αρνητικά σε ένα τέτοιο αίτημα. Εγώ αυτό που θέλω σαν νομικός είναι μία λέξη σέρτα, δηλαδή μία, ε, μία νομοθεσία η οποία να μην αφήνει κανένα περιθώριο διαφορετικής ερμηνείας. Θέλω σαφήνεια νόμου. Επίσης, ε, συχνά αναρωτιέμαι τι θέλουν να κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες με όλα αυτά τα δεδομένα. Αν είχατε διαβάσει τη συμφωνία FTP θα ξέρετε ότι ένα άρθρο αναφέρει ότι απαγορεύεται να γίνεται ε, αυτό που στα αγγλικά ονομάζεται data mining. Αλλά όταν κάποιος ε, κάθε μέρα ας πούμε δέχεται ε, αυτά τα ε, δεδομένα χίδιν οπωσδήποτε θα πρέπει να τα αντιμετωπίσει μέσω της διαδικασίας data mining. Και το ίδιο διαπιστώνω μιλώντας και με την ε, συνάδελφο που είναι υπεύθυνη από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Η κυρία Σίπολ με ρώτησε εάν συζητήθηκε η συμφωνία αυτή με την Επίτροπο Μάλστρομ. Όχι. Όχι, δεν δεχτήκαμε κανένα αίτημα από πλευρά της Επιτρόπου ε, να συζητήσουμε και δεν είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε για το θέμα αυτό και για τα πορίσματα της μελέτης μας. Ε, εγώ προσωπικά απέστειλα επιστολή σε σχέση και με την σύγκρουση ε, συμφερόντων ε, η οποία βαρύνει δύο συναδέλφους αλλά για την ώρα δεν ε, έλαβα απάντηση για την επιστολή μου αυτή. Ίσως για να οδηγηθούμε λίγο και προς το τέλος η συμφωνία TFTP, όπως και η ιστοσελίδα της Κομισιόν έχουν την συμφωνία αυτή ε, σεβόμενοι πάντως την ε, προστασία των ε, στοιχείων και δεδομένων εμπιστευτικού χαρακτήρα των πολιτών. Και πρέπει να σας πω πάντως ότι η συμφωνία αυτή δεν κάνει το ίδιο, δηλαδή δεν σέβεται την προστασία και την εμπιστευτικότητα των προσωπικών στοιχείων των πολιτών. Ευχαριστώ πολύ. Είπατε, αν κατάλαβα καλά, ότι αυτή η συμφωνία ε, δεν ε, ε, σέβεται την εμπιστευτικότητα. Ναι, εννοείται, φαντάζομαι, την προστασία των ιδιωτικών εμπιστευτικών δεδομένων. Συνάδελφοι, έχουμε πέντε λεπτά πριν ξεκινήσει η εξέταση του επομένου σημείου. Να σταματήσουμε λοιπόν, να διακόψουμε για λίγα λεπτά και θα δώσω ξανά την Προεδρία στην κυρία Μπάουερ.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 Uh, uh, uh, Καλημέρα σας ξανά. Φτάσαμε στο σημείο 9 και 10 της ημερησίας διατάξεως, τα οποία θα συζητήσουμε από κοινού. Ο κύριος ε, Δίας Δεμέρα είναι ο εισηγητής μας. Ε, ταυτόχρονα θα κάνουμε και ανταλλαγή απόψεων με τον κύριο Μπάμφη, διευθυντή της ε, ΣΕΠΟΛ και τον κύριο Ρόμπ Βενράιτ, διευθυντή της Ευρωπόλ, σχετικά με την πρόταση όσον αφορά τη συγχώνευση Europol και ε, ΣΕΠΟΛ. Ζητούμε συγγνώμη εκ των προτέρων που δεν είναι πολλοί οι βουλευτές, αλλά πρέπει να σας πω ότι αυτή τη στιγμή λαμβάνει η χώρα μια σημαντική ψηφοφορία στην Επιτροπή ΚΡΙΜ ε, και γι' αυτό πολλοί βουλευτές είναι εκεί. Λοιπόν, ε, ε, πρέπει να συζητήσουμε πάντως τα θέματα αυτά, διότι επιγόντως πρέπει να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις ε, πριν τις ευρωπαϊκές ε, εκλογές. Ε, γι' αυτό λοιπόν έχουμε τώρα την πρώτη συζήτηση και για το πρώτο θέμα που είναι η συνεργασία σχετικά με την βουλή του νόμου και την κατάρτιση, την Europol και κατάργηση κάποιων αποφάσεων και μετά την συζήτηση που αφορά και την ΣΕΠΟΛ. Ε, πρώτα θα ακούσουμε την Κομισιόν για μια σύντομη παρουσίαση της πρότασης. Μετά θα ζητήσω από τον εισηγητή κύριο Ντίας Δεμέρα να πάρει το λόγο και να παρουσιάσει τις δικές του απόψεις επί της προτάσεως. Και μετά θα δώσω το λόγο στους ε, καλεσμένους μας. Πρώτα απ' όλα ε, στον κύριο Ζων Μάχονη και μετά στον κύριο Φίντεν Φάνη ε, αντίστοιχα ε, διευθυντή ε, του Συμβουλίου της Europol και της ΣΕΠΟΛ έτσι ώστε να μας μιλήσουν και για την πρόταση αλλά και για την πρόταση συγχώνευσης Europol Επολ, και μετά θα ξεκινήσει η συζήτηση με τους βουλευτές που ελπίζω να είναι πολυπληθέστεροι πλέον. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να ζητήσω από την Κομισιόν να πάρει το λόγο και να παρουσιάσει τις προτάσεις της. Ποιος είναι εκπρόσωπος εδώ της Κομισιόν, η κυρία Μίτσι. Βλέπω και τον κύριο Μοσαβίζη. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Κοινοβουλίου, κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα ε, να σας διαβιβάσω την, ε, ε, τις Τη λύπη του κυρίου Πριβέρου που δεν μπορούσε να είναι εδώ δυστυχώς και θα ήθελα να τον δικαιολογήσετε γι' αυτό. Έχουν ε, υποβληθεί ήδη και από την ε, κυρία Μάλστρομ κάποιες απόψεις της Κομισιόν ενώπιον της Επιτροπής σας Λίμπε. Ε, με την ε, εφαρμογή της συνθήκης της ε, Λισαβόνας το θέμα της Europol έχει πάρει ιδιαίτερη σημασία. Η κυρία Μάλστρομ κατέστησε σαφές ήδη στις αρχές του 2010 λαμβάνοντας υπόψη και την ευαισθησία του Κοινοβουλίου ότι θα πρέπει με συναπόφαση να εγκριθεί η πρόταση αυτή, η οποία με τη σειρά θα πρέπει να προετοιμαστεί με μεγάλη προσοχή. Ε, λαμβάνοντας υπόψη και το input ε, πολλών φορέων αλλά κυρίως και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ξεκίνησε λοιπόν ο διάλογος ε, με τους οποίους συμμετέχουν και μέλη της Επιτροπής σας εδώ και εκπρόσωποι των κρατών μελών του EDPS καθώς επίσης και εμπειρογνώμονες και μέλη των διοικητικών οργάνων των δύο ε, οργανισμών. Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα στοιχεία, ε, εξ αρχής ε, στόχος της Κομισιόν ήταν να δημιουργήσει μια, έναν οργανισμό ή μια υπηρεσία η οποία θα είναι πιο αποτελεσματική, θα δίνει καλύτερα αποτελέσματα και σε επίπεδο λογοδοσία θα είναι καλύτερη. Ε, για πρώτη φορά μάλιστα ε, εμπλέκονται τα Εθνικά Κοινοβούλια στη διαδικασία αυτή. Θεωρούμε ότι για να μπορέσει να υπάρξει σωστή επιβολή του νόμου θα πρέπει και η κατάργηση να είναι σωστή, η κατάρτιση να είναι σωστή και ο βαθμός λογοδοσίας να είναι ικανοποιητικός. Τα ίδια τα κοινοβούλια βεβαίω θα πρέπει να αποφασίσουν και όχι οι Κομισιόν. Και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα Εθνικά Κοινοβούλια σαφώ έχουν σημαντικό ρόλο να παίξουν ε, στην διασφάλιση τη σωστή και αποτελεσματική εργασία ε, του ε, οργανισμού, κυρίω δε σε σχέση με τα όσα προβλέπονται για τη λειτουργία αυτή στο καταστατικό. Στις νέες διαδικασίες προβλέπεται και αξιολόγηση εκ των προτέρων εξάντε Προτείναμε λοιπόν το ε, ε, Διοικητικό Συμβούλιο ε, του, της Ευρωπόλ να υποβάλει πολυετές πρόγραμμα έτσι ώστε να μπορεί να λαμβάνει η χώρα στρατηγική συζήτηση για τους προσανατολισμούς που θα πρέπει να ακολουθήσει ο οργανισμός. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα Εθνικά Κοινοβούλια θα λαμβάνουν όλες τις θέσεις της Europol που δεν είναι διαβαθμισμένες καθώς επίσης και μια στρατηγική ανάλυση σε σχέση με τους στόχους της Ευρωπόλ. Και τέλος ε, και τα αποτελέσματα των μελετών που έχει ε, ξεκινήσει η Europol. Οποτεδήποτε χρειάζεται ε, θα δίνεται πιο ενδελεχής η εικόνα στο Κοινοβούλιο που θα έχει την δυνατότητα με τη σειρά του να ζητάει πρόσβαση σε διαβαθμισμένα έγγραφα που έχει η Europol στη διάθεσή της. Ε, θα υπάρξει μια διευθέτηση εργασιών μεταξύ του Κοινοβουλίου και της Europol. Όσον αφορά τώρα την εξπόστα εκ των υστέρων εποπτεία και το Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα Εθνικά Κοινοβούλια ε, θα έχουν ε, τα πρακτικά καθώς επίσης και όλες τις αξιολογήσεις και την έκβαση των αξιολογήσεων που κάνει η Κομισιόν. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επίσης θα έχει την δυνατότητα να, όπως και κάθε άλλο ε, διακοινοβουλευτικό φόρουμ, θα έχουν την δυνατότητα, λέγω, να εγκαλούν τον πρόεδρο, διευθυντή ή διευθύνοντα σύμβουλο ε, της Ευρωπόλ. Όσον αφορά τώρα το δεύτερο στόχο μας, ε, δηλαδή να γίνει πιο αποτελεσματική η Ευρωπόλ στην στήριξη των κρατών για την καταπολέμηση των εγκλημάτων. Ε, και ε, των εγκληματικών δραστηριοτήτων. Ε, σε αυτό χρειάζεται μεγαλύτερη στήριξη η Ευρωπόλ. Θέλει περισσότερα δεδομένα, στοιχεία, ανάλυση εγκληματικών διεργασιών κτλ. Διασφαλίζεται, συγγνώμη, αποσαφηνίζεται από την Κομισιόν και το input που θα πρέπει να δίνουν τα κράτη-μέλη προς την Ευρωπόλ. Επίσης, την χρηματοδοτική στήριξη για μεμονωμένες μελέτες όπως αυτά ας πούμε, που λαμβάνουν χώρα τούτη τη στιγμή ε, στον τομέα της παραχάραξης. Επίσης, ε, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα λαμβάνουν ετήσια ε, ανάλυση των στοιχείων που έχουν λάβει από τα κράτη-μέλη. Όμως δεν αρκούν τα ίδια τα δεδομένα. Γι' αυτό το λόγο η πρόταση ε, θέλει να ε, οθήσει ε, και να προωθήσει την αναλυτική ικανότητα της Ευρωπόλ στα πλαίσια μιας βάση δεδομένων που δεν θα είναι προδιαγραμμένη εκ των προτέρων και βεβαίως η διαχείριση όλων των στοιχείων, οι πηγές των πληροφοριών θα είναι καλά προγραμματισμένες. Ε, υπάρχουν ε, κατηγορίες ε, στοιχείων προσωπικών και μη που οπωσδήποτε θα συλλέγονται για συγκεκριμένους στόχους. Ε, θα πρέπει ε, με τον τρόπο αυτό η Ευρωπόλ ε, να καταφέρει να δώσει μια καλύτερη αποτελεσματική, αποτελεσματικότερη εικόνα όσον αφορά τα ίδια τα δεδομένα, την ταξινόμησή τους, τη διαχείρισή τους, τον τρόπο λειτουργίας των εγκληματιών κτλ. Ε, όσον αφορά την προστασία των ε, στοιχείων των πολιτών. Ε, στην πρόταση μας υπάρχει μια πάρα πολύ ισχυρή προστασία των προσωπικών δεδομένων. Ε, χρειαζόμαστε μεγαλύτερη διαφάνεια καθώς επίσης και σαφήνεια νόμου και για πρώτη φορά ε, έχουμε τόσο συγκεκριμένους ε, τόσο συγκεκριμένες αρχές οι οποίες βρίσκονται σε ένα και μόνο νομικό εργαλείο. Ε, η ε, απόφαση 45 του 2001 είναι ε, αυτή τη στιγμή τροποποιημένη και επίσης λαμβάνοντας υπόψη και την ιδιαιτερότητα της προστασίας των δεδομένων στα πλαίσια της επιβολής του νόμου δίνεται ένα αυτόνομο καθεστώς κατά αυτή την έννοια στην Ευρωπόλ θα υπάρχει και δυνατότητα εξωτερικής επόπτευσης. Ε, το ε, EDPS καλύπτει όλα τα στοιχεία ανεξαρτησίας τα οποία έχει ορίσει ε, το δικαστήριο. Ταυτοχρόνως δε έχει όλα τα στοιχεία και τις δυνατότητες αρμοδιότητες για να μπορέσει να λειτουργήσει σωστά. Ε, τα προσωπικά στοιχεία τα οποία ε, κρατάει η Ευρωπόλ ε, βασίζονται στο σύστημα διπλού hit. Δηλαδή, ενδεχομένως μπορεί να υπάρξει ένα πρώτο hit όσον αφορά την, ε, ε, όσον αφορά την ταύτιση των στοιχείων, αλλά μονάχα εάν υπάρχει ένα δεύτερο hit, δηλαδή μια δεύτερη διαδικασία που θα καλύπτει περαιτέρω εχέγγυα, μόνο τότε θα υπάρξει η ανταπόκριση η Ευρωπόλ είναι ε, υποχρεωμένη μετά από αίτημα του ενδιαφερόμενου ε, να του δώσει όλα τα στοιχεία του ΙΤΙΣ που έχει στη διάθεσή της ε, η Ευρωπόλ και έχει δυνατότητα να έχει πρόσβαση στοιχεία αυτά. Οποιοςδήποτε μπορεί να ζητήσει αποζημίωση από την Ευρωπόλ για εσφαλμένη χρήση των στοιχείων, των δεδομένων της και η προσφυγή μπορεί να λάβει χώρα στην χώρα ε, στην οποία ε, το αδίκημα έχει λάβει χώρα. Ε, όσον αφορά την προστασία θυμάτων, μαρτύρων, ανηλίκων, είναι σαφής και απαγορεύεται η χρήση των δεδομένων τους παρά σε κάποιες ειδικές περιπτώσεις. Δεν ε, επίσης ε, ε, δεν είναι δυνατόν να μεταφέρονται στοιχεία τα οποία ονομάζομαι γενικά ευαίσθητα και τα οποία αφορούν την θρησκεία, την εθνότητα, τις σεξουαλικές προτιμήσεις κτλ. Ε, στρατηγικού ενδιαφέροντος και τεχνικού χαρακτήρα στοιχεία μπορούν να ανταλλάσσονται με τρίτες χώρες, αλλά τα προσωπικά στοιχεία μεταφέρονται σε τρίτες χώρες μονάχα ε, επί τη βάση διεθνών ε, συμφωνιών που έχει υπογράψει με τις χώρες αυτές η Ευρωπαϊκή Ένωση ή μετά από ειδική συμφωνία με την Κομισιόν ή βάση προϋπάρχουσας συμφωνίας μεταξύ Europol και ε, τρίτης χώρας και εν πάση περιπτώσει οι αποφάσεις θα λαμβάνονται ε, σε ε, αναπερίπτωση από τον Διευθυντή της Europol. Όσον αφορά την βελτίωση της αποτελεσματικότητας η κατάρτιση είναι πάρα πολύ σημαντική, η κατάρτιση των αξιωματούχων της επιβολής του νόμου. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να ενισχυθεί η αστυνομική συνεργασία αφενός και η, κατάργηση, συγγνώμη, και η κατάρτιση και η εκπαίδευση αφετέρου. Με τον τρόπο αυτό η Ευρωπόλ ε, θα μπορέσει ε, να αντιμετωπίσει τις ε, απαιτήσεις της Κομισιόν όσον αφορά την επιβολή του νόμου και την κατάρτιση έτσι όπως ε, αυτά αναφέρονται στους ε, κανονισμούς. Όσον αφορά την Αστυνομική Ακαδημία, η Ευρωπόλ ε, θα στηρίξει, θα συντονίσει, θα προωθήσει την κατάρτιση των αξιωματούχων της επιβολής του νόμου σε κάθε επίπεδο και όχι μονάχα των υψηλόβων αξιωματούχων όπως συμβαίνει τώρα για την ε, ε, Κομισιόν. Ε, η Κομισιόν θεωρεί ότι όλοι όσοι ασχολούνται με την επιβολή του νόμου, ανεξαρτήτως βαθμίδας, θα πρέπει να έχουν την, τις ίδιες δυνατότητες κατάρτισης. Είτε μιλάμε για αστυνομικούς που μόλις έχουν βγει από την Ακαδημία της Αστυνομίας, είτε μιλάμε για τελωνιακούς επαλλήλους. Παντού η διαστηνοριακή συνεργασία είναι πάρα πολύ σημαντική για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος. Επίσης ε, θέλουμε να παράσχουμε εξειδικευμένη κατάρτιση όσον αφορά οι ιδιαίτερες μορφές ε, του οργανωμένου εγκλήματος, ε, ξέπλυμα χρήματος, τράφικινγκ κτλ. Τέλος, και σε σχέση με τη διακυβέρνηση και βεβαίως και όσον αφορά τη λογοδοσία, η ε, ε, Ευρωπόλ είναι ε, μία από τις πρώτες υπηρεσίες οι οποίες θα λειτουργήσουν με βάση της αποκεντρωμένης διοίκησης που αποφασίστηκε πέρσι το καλοκαίρι από την Κομισιόν, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Να σας πω και κάποια στοιχεία η σύσταση, η σύνθεση μάλλον της, του Διοικητικού Συμβουλίου έχει αλλάξει έτσι ώστε να είναι σαφέστερη η εικόνα της Europol ως εργαλείο επιβολής του νόμου η διοικητική αυτή επιτροπή θα συνεπικουρείται από ε, εμπειρογνώμονες έτσι ώστε να διασφαλιστούν τα μεγαλύτερα δυνατά επίπεδα ε, κατάρτισης τεχνογνωσίας και αποτελεσματικότητας. Μέχρι τώρα το, μόνο το Συμβούλιο έχει τη δυνατότητα να ορίσει ε, τους διευθυντές και πρόεδρους της Europol. Πλέον αυτό θα γίνεται από το Management Board με στόχο βεβαίως και, και ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να καλέσει τους ε, υποψηφίους ε, για τη θέση του Αντιπροέδρου και του Προέδρου ενώπιόν του έτσι ώστε να συζητήσει μαζί τους και αυτό στα πλαίσια της μεγαλύτερης διαφάνειας και της του καλύτερου βαθμού λογοδοσίας. Ευχαριστώ πολύ. Έχω... Λιγότερο από μία ώρα για να συζητήσουμε με τα μέλη του πάνελ και βέβαια τους βουλευτές να ακούσουμε όλες τις πανεβάσεις. Γι' αυτό θα παρακαλέσω να είναι ο καθένας το δυνατόν πιο συνοπτικός. Θα καλέσω τώρα τον κύριο Δίας Δεμέρα, τον εισηγητή, να λάβει το λόγο για τα αρχικά του σχόλια. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Όμως, πρωτού λάβω το λόγο, θέλω να σας προτείνω αν είναι δυνατόν, να ακούσουμε πρώτα την άποψη του Συμβουλίου. Να ρωτήσουμε το Συμβούλιο λοιπόν, εάν θέλουν να μιλήσει πρώτο. Ποιος το εκπροσωπεί εδώ. Θέλετε να λάβετε το λόγο πρώτος, για να σύντομο σχόλιο. Ευχαριστώ. Εκ μέρου ε, τη Προεδρία θα ήθελα να πω ότι λάβαμε επιστολή από τον ε, Πρόεδρο τη Επιτροπή σα. Έλαβε ο Πρόεδρό μα δηλαδή. Μελετάει τι προτάσει, θα απαντήσει σύντομα. Αύριο στη συνεδρίαση ΚΑΤΣ. Και φαντάζομαι και στο Συμβούλιο των, της Δικαιοσύνης και Εσωτερικών θα συζητηθεί τον Ιούνιο. Αλλά μέχρι τώρα δεν έχω τίποτα άλλο να πω. Κατάλαβα. Άρα θα επανέλθετε έτσι, δηλαδή αύριο και τον Ιούνιο με το Συμβούλιο. Ευχαριστώ πολύ και εφόσον δεν έχουμε άλλα στοιχεία από το Συμβούλιο, ας λάβει το λόγο η Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα κάνω κάποια σύντομα εισαγωγικά σχόλια. Και το πρώτο που θέλω να πω είναι ότι λυπούμε που η μετάφραση του νομοθετικού κειμένου στις γλώσσες Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν έτοιμη χθε το απόγευμα και αυτό μόνο κατόπιν ετήματος και υπό τις συνθήκε αυτές καταλαβαίνετε δεν μπορεί κανεί να εργαστεί με σοβαρότητα. Εξκουσάει τον πετίτα βέβαια και έχουμε εργαστεί, έχουμε εργαστεί πολύ καιρό για το ενδεχόμενο δρομολόγηση αυτή τη τόσο απαραίτητη νομοθετική πρωτοβουλία. Μιλάμε για έναν οργανισμό, για ένα ε, γραφείο Ευρωπαϊκής Αστυνομίας, όπως είναι Ευρωπόλ που δεν μπορούσε από νομικής πλευράς να ε, υπάγεται σε απόφαση του Συμβουλίου. Γιατί αυτό την καθιστούσε εύθραυστη από νομικής πλευράς. Επομένως, στηρίζουμε αυτήν την νομοθετική όθηση που σήμερα αρχίζει να δίνεται ώστε τελικά η Europol, η Ευρωπόλ να έχει την νομική, το νομικό καθεστώς που της αρμόζει. ένα κοινοτικό δηλαδή οργανισμό, κανονισμού. Θέλω να ευχαριστήσω την Κομισιόν για την παρουσίαση που μας έκανε. Και πρωτού επισέλθω σε άλλα θέματα, θα ήθελα να πω ότι ο κανονισμός έχει 14 κεφάλαια. Η νομοθετική πρόταση έχει 14 κεφάλαια και 79 άρθρα. Ένα νεωτερικό στοιχείο που είναι βέβαια αμφιλεγόμενο και πολύπλοκο είναι στο κεφάλαιο 3, το θέμα της συγχώνευσης συγκεκριμένα. Το θέμα της συγχώνευσης ε, θα συζητηθεί ευρύτερα στο σημείο 10 της ε, συνεδρίασής μας. Όπως και να έχει όμως, θέλω να πω το εξής. Το νομοθετικό κείμενο μπορεί να βελτιωθεί σε ό,τι αφορά το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εκτελεστική Επιτροπή. Κάτι νέο που δεν ήταν στην πρόταση του Συμβουλίου. Θα πρέπει όμως να πούμε και κάτι σε σχέση με τον ορισμό, την εκλογή του Διευθυντή. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπως είναι φυσικό, δεν θα παρέμβει στην διαδικασία επιλογής που δυνάμει της απόφασης του Συμβουλίου ήταν μία πρόταση με τρία ονόματα το Συμβουλίο, το Διοικητικό. Και με βάση τις προτάσεις της Κομισιόν θα έχουμε μία πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου. Δεν έχουμε να πούμε κάτι αρχικά, αλλά σε ό,τι αφορά το ρόλο του Κοινοβουλίου στην όλη διαδικασία, έχουμε να πούμε κάτι. Και συμπεριλαμβάνεται εδώ και η διαδικασία της επιλογής του ορισμού μάλλον του διευθυντή και όχι στη διαδικασία της επιλογής, στη διαδικασία του ορισμού. Και έχουμε και το θέμα του κοινοβουλευτικού ελέγχου. Μιλάμε εδώ και καιρό για τον κοινοβουλευτικό έλεγχο και πρέπει το νομοθετικό κείμενο να βελτιωθεί. Η νομοθετική πρόταση πρέπει να γίνει καλύτερη στο σκέλος αυτό. Γιατί, Γιατί θέλουμε να είναι αποτελεσματικός αυτός ο κοινοβουλευτικός έλεγχος και όχι κατά ανάγκη σε σχέση με αυτό που η κυρία Μίτσι, εξάντε και εξ έλεγχος. Όχι. Και αυτό βέβαια, αλλά θα πρέπει να μελετήσουμε τον ακριβή τύπο, την ακριβή φόλμορα που θα επιτρέψει την ε, εφαρμογή αυτού του ελέγχου και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και από τα Εθνικά Κοινοβούλια. Θα πρέπει να αξιολογήσουμε λοιπόν ε, το θέμα αυτό γίνει στο δυνατόν πιο αποτελεσματικό ο έλεγχο. Επίση, επεξεργασία των πληροφοριών, που είναι και η πεμπτουσία τη Europol ουσιαστικά. Λαμβάνει πληροφορίε, επομένω, με έναν οργανισμό, με έναν κανονισμό, θα είναι πιο ομαλή η ροή των πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών και της Europol και βέβαια πρέπει να έχουμε υπόψη μας και την ανάγκη ασφάλειας. Πρέπει λοιπόν να υπάρχουν πολλά και καλά χέγια. Φυσικά πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη προστασία και ενίσχυση ε, του καθεστώτος προστασίας δεδομένου προσωπικού χαρακτήρα. Για πρώτη φορά σε με αυτό που προβλεπόταν στην πρόταση του Συμβουλίου, εδώ ενισχύεται και ο ρόλος του Ευρωπαίου Πόπτη. Πριν αξιολογήσω τα σχόλια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θέλω να πω κάτι ακόμη. Είμαι απόλυτα στη διάθεση των συναδέλφων οι οποίοι θα οριστούν σκιώδη ε, σκιώδεις εισηγητές. Είμαι απόλυτα στη διάθεσή του το λέω και πάλι. Και βέβαια θα είμαι ε, διατεθμένος να οργανώσω όσο, όσες συναντήσεις χρειαστεί για να γεφυρώσουμε τις διαφορές μας, αν υπάρχουν. Να σας πω και κάτι για το χρονοδιάγραμμα. Εμείς θα πρέπει να έχουμε ολοκληρώσει τις εργασίες μας ε, σίγουρα πριν λήξει η τρέχουσα κοινοβουλευτική περίοδος. Παραλαμβάνω, θα εργαστώ, θα αφοσιωθώ ε, στην έκθεση αυτή. Και τώρα να απαντήσω στην κυρία Μίτσι, στη Βικτόρια. Και σε όλους εσάς θέλω να πω ότι είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος που εκπροσωπεί η Βικτόρια την Κομισιόν γιατί είναι πάρα πολύ καλή επαγγελματία, γνωρίζει σε βάθος αυτά τα θέματα που μας απασχολούν, γνωρίζει σε βάθος την Ευρωπόλ και έχω το προνόμιο να έχω συνεργαστεί μαζί της πριν πολύ καιρό βέβαια. Έρχομαι τώρα στην ουσία της παρουσίας της Κομισιόν. Νομικό πλαίσιο, πρώτα απ' όλα. Δεν το συζητάω ε, επί της αρχής, αλλά επειδή θα ακούσουμε και τους εκπροσώπους των ε, οργανισμών και της Αστυνομικής Ακαδημίας ε, όλες ιδιαίτερος, θέλω να θέσω υπόψη στο θέμα του άρθρου 87 και του άρθρου 88. Τη σκοπιμότητα των δύο άρθρων αυτών. Είναι επίμαχο το θέμα. Το νομικό πλαίσιο όμως πρέπει να το συζητήσουμε. Θα μας απασχολήσει. Συμφωνώ με την κυρία Μίτση ως προς τη σημασία που έχει να δώσουμε νέα πνοή στον κοινοβουλευτικό έλεγχο, να τον αναζωογονήσουμε. Και σε ό,τι αφορά το δεύτερο στόχο που είναι η αποτελεσματική καταπολέμηση του εγκλήματος και η καλύτερη συνεργασία με τα κράτη-μέλη. Πράγματι, είναι απολύτως αναγκαίο αυτό για να ενισχυθεί και η δομή της Europol. Σίγουρα πρέπει να έχουμε μια πιο ισχυρή από νομικής πλευράς δομή σε ό,τι αφορά την συλλογή, επεξεργασία, προστασία και ε, διαβάθμιση στοιχείων προσωπικού χαρακτήρα. Φυσικά πρέπει να δημιουργήσουμε ένα σύστημα προστασίας δεδομένων που θα είναι αποτελεσματικό, θα είναι συμπαγές και θα προσφέρει εγγύησεις. σε ό,τι την κατάρτιση, την εκπαίδευση. Καλύτερα ίσως να αναβάλω ε, για μια μεταγενέστερη συζήτηση τα σχόλια μου πάνω σε αυτό, γιατί πρώτα θα ήθελα να ακούσω τι θα πούν η ε, Ευρωπόλ, η ΣΕΠΟΛ και τα ΔΕΛΤΑ ΣΥΓΜΑ των οργανισμών αυτών. Προκαταβολικά όμως μπορώ να πω ότι προσωπικά εγγράφως έχω δηλώσει ότι ήμουν αντίθετος με την συγχώνευση. Ήμουν αντίθετος, πέραν αυτού όμως είμαι σε θέση και να μιλήσω και να ακούσω και να ε, δείξω και κάποια ευελιξία. Με στόχο βέβαια να ενισχυθεί η καταστατική ρυθμιστική λειτουργία των δύο αυτών οργανισμών. Αυτά έχω να σας πω για την Επιτροπή. Για το Συμβούλιο δεν έχω να πω τίποτα. Απλά εκφράζω τη λύπη μου για τα τόσα λίγα που μας είπε το Συμβούλιο. Τώρα, το ότι έρχεται το Συμβούλιο και μας λέει ότι θα απαντήσει στην επιστολή του κυρίου Λόπεθ Αγιλάρ και είτε τώρα είτε στο Συμβούλιο Δικαιοσύνης Εσωτερικών τον Ιούνιο θα αποφανθεί και θα μας πει αυτό πραγματικά συνιστά παινία, σημαντική παινία ε, ενημέρωση πληροφόρησης και αυτό είναι λυπηρό από μόνο του. Ξέρουμε ότι θα συζητηθεί ένα θέμα αύριο και θα συζητηθεί και στο Συμβούλιο Δικαιοσύνης Εσωτερικών. Θα ακούσουμε τους εκπροσώπους ε, Ευρώπολη και ΣΕΠΟΛ και όλα αυτά που θα μας πούν θα έπρεπε να τα είχαν συζητήσει τα, τα κράτη. Τα κράτη βέβαια έχουν λάβει τις σχετικές προτάσεις και πληροφορίες. 16 κράτη-μέλη έχουν εκφραστεί ότι θα το συζητήσουν αύριο ή τον Ιούνιο, εντάξει. Αλλά αυτό που θέλω να πω στο Συμβούλιο είναι ότι πρέπει να ασχοληθούν σοβαρά με το νομοθετικό αυτό καθήκον. Δεν μπορούν να λένε θα δούμε ίσως αύριο κάτι πιο συγκεκριμένο περιμένω. Αυτά είχα να πω. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ για την πολύ σαφή τοποθέτηση στα θέματα αυτά. Είναι σημαντικό να ξεκινήσει η συζήτηση και θα ζητήσω πρώτα τον κύριο Ομαχώνη, που είναι ο πρόεδρος του, του Συμβουλίου της Europol να λάβει το λόγο. Παρακαλώ, για πέντε λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Και ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να συζητήσουμε την δυνατότητα, την προοπτική αυτή συγχώνευσης της Europol με τη ΣΥΠΟΛ. Το Δικαιωτικό Συμβούλιο σε πρόσφατες συνεδριάσεις του συζήτησε ε, εν συντομία τα θέματα αυτά, αλλά δεν έχει μπορέσει να συζητήσει διεξοδικά και να δει τα στοιχεία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ως εκ τούτου για να λάβει απόφαση με τα λογογνώσεως θα πρέπει να λάβει περισσότερα στοιχεία και να ολοκληρώσει και τη συνεδρίαση του 22 Μαΐου στη Χάγη για να έχουν τη δυνατότητα και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να συστήσουν τα διάφορα ζητήματα. Μετά τη δημοσίευση στις 27 Μαρτίου του 2013 της πρότασης αυτής, εγώ εξέτασα το θέμα και ζήτησα από το Διοικητικό Γραμματεία του Διοικητικού Συμβουλίου να ξεκινήσει μια γραπτή διαδικασία ε, για να εξετάσει τα υπέρ και τα κατά αυτή τη προτινόμενη συγχώνευσης. 18 ήταν οι φορέ που λάβαμε. Η κυρία θέση του Διοικητικού Συμβουλίου δεν υποστηρίζει την προτινόμενη συγχώνευση μεταξύ Europol και ΣΥΠΟΛ και θα ήθελα να σας δώσω τα κύρια στοιχεία αυτών των, ε, τους κύριους λόγους που προβλήθηκαν. Οι δύο υπηρεσίε καταρχάς έχουν ε, θεμελιωδώς διαφορετικές εντολές, δεν παρουσιάζουν επικάλυψη. Στι εντολές τους. Η ΣΥΠΟΛ έχει δραστηριότητες πολύ διαφορετικές και πέραν αυτών της Europol για την ε, πρόληψη, τη διαχείριση των συνόρων, την επιβολή της τάξης και την ενημέρωση των νεαρών αστυνομικών για τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα πέραν των στόχων λοιπόν της Europol και την διασφάλιση της ε, κατάρτισης των αστυνομικών δυνάμεων σε περιπτώσεις μη στρατιωτικό ή κρίσεως. Όλα αυτά λοιπόν θα έπρεπε να τα αναλάβει σε περίπτωση συγχώνευσης η Europol. Υπάρχουν κάποια παραδείγματα ε, των στόχων και του λόγου ύπαρξης της ε, ΣΥΠΟΛ που εξετάστηκαν που, κρίνεται ότι ξεπερνούν σε μεγάλο βαθμό το ρόλο και τα καθήκοντα της Europol όπως ορίζεται στο άρθρο 68 της συνθήκης. που έχει να κάνει περισσότερο με τη συνεργασία μεταξύ αστυνομικών αρχών για την καταπολέμηση τη σοβαρή εγκληματικότητα, τη τρομοκρατία, του οργανωσμένου εγκλήματο, μέσα από την ε, Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και το πλαίσιο που ορίζει αυτή. Ω εκ τούτου, εάν αναλάβει τα καθήκοντα τη ε, ΣΥΠΟΛ, Europol, ενδέχεται να ε, βρεθεί σε αδυναμία να επιτελέσει το βασικό της καθήκον σε μια, περίπτωση, σε μια περίοδο που προσπαθεί να θεσπίσει το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Καταπολέμηση του Κύβερνο Εγκλήματος. Η κατάρτιση επίσης ε, μπορεί να καταστεί ε, δευτερεύουσα σημασία καθήκων και τελικά να υποβαθμιστεί. Τα ε, καθήκοντα των δύο αυτών υπηρεσιών συνεπάγονται, απαιτούν ειδικέ ικανότητες και η καταπολέμηση της ε, τρομοκρατίας αλλά και η κατάρτιση των αστυνομικών δυνάμεων ε, πρέπει να παραμείνουν στα χέρια διαφορετικών ε, θεσμικών, διαφορετικών οργάνων, διαφορετικών οργανώσεων. Επίσης, με βάση αποφάσεις του Βουλίου του Κοινοβουλίου, αναφέρεται ότι μπορεί να γίνει συγχώνευση όταν παρουσιάζονται στοιχεία ε, επικάλυψης στα καθήκοντα των φορέων ή οργανισμών, πράγμα το οποίο δεν ισχύει με τη ΣΥΠΟΛ και τη Europol. Δεν βλέπουμε πώς θα μπορούσαν δηλαδή, να λειτουργήσουν σε μια ευρύτερη ε, δομή που θα μπορούσε να προκύψει από μια συγχώνευση. Επίσης από, τους, ε, από τις απαντήσεις που λάβαμε εκφράστηκαν πολλές ε, αμφιβολίες για το κατά πόσον θα προκύψει οικονομικό όφελος ή εξοικονόμηση πόρων δεν είναι αρκετά λεπτομερή ε, στο στοιχείο, στο σημείο αυτό η πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και δεν λαμβάνεται υπόψη το γεγονό ότι μπορεί με την συγχώνευση αυτή να χρειαστούν διαφορετικές και νέε, ε, διαφορετικοί και νέοι ανθρώπινοι αλλά και ηλικοί πόροι. Μετά τη συγχώνευση λοιπόν θα χρειαστούν πόροι οι οποίοι θα θέσουν σε κίνδυνο την ορθή επιτέλεση του έργου τόσο της Ήπολος όσο και της Πυροπόλου. Η ΣΥΠΟΛ εργάζεται, συνεργάζεται πολύ καλά με την Europol, αλλά και με τα κράτη-μέλη και με άλλους οργανισμούς και φορείς Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η συγχώνευση αυτή μπορεί να μειώσει την ορατότητα της ΣΥΠΟΛ, γιατί θα ευθυγραμμιστεί αναγκαστικά αυτή η, εταιρεία, η επιχείρηση στις ε, εργασίες κατά πολέμηση του εγκλήματος και βέβαια και η συνεργασία με τα κράτη-μέλη όπως προς την καθηδήγηση των εργασιών της για την καταπολέμηση του εγκλήματος και την υποβολία της τάξης και άλλες ευρωπαϊκές ε, οργανώσεις ή φορείς έχουν συνεργαστεί με την ΣΥΠΟΛ και την Europol όπως είπαμε ε, ειδικότερα στο θέμα της συνεργασίας για την ε, επιβολή του νόμου και όχι την κατάρτιση όσον αφορά την Europol και άρα όπως είπαμε θα πρέπει να συνεχίσει να δραματίζει τον ουσιώδη ρόλο της Europol στην καταπολέμηση του εγκλήματος. Μένει το ερώτημα λοιπόν, γιατί να μην περιλάβει και την Frontex, εφόσον είναι και αυτή ένα συνεργαζόμενο οργανισμό, αυτή η συγχώνευση. Η νέα εντολή δεν θα είναι σύμφωνη με το άρθρο 88 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ορίζει το Συμβούλιο με βάση την νομοθεσία και τακτική νομοθετική διαδικασία θα ορίσει τον τρόπο λειτουργίας, το, τα καθήκοντα, την εντολή και ε, τη δομή της Europol. Αυτό δεν προβλέπεται από τη συνθήκη, δηλαδή το να επιβληθούν και νέα καθήκοντα στην ε, Europol. Μπορεί κάπου όταν υπάρχουν συνεργατικές σχέσεις, όταν υπάρχουν παράλληλες ε, ε, αρμοδιότητες μεταξύ ε, φορέων και υπηρεσιών έχει νόημα μια συγχώνευση, αλλά δεν φαίνεται να έχει κανένα θετικό ε, αποτέλεσμα να παραγάγει στην προκείμενη περίπτωση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν έχει δώσει μια ενημέρωση για την προτινόμενη νομοθεσία, για τον προτινόμενο κανονισμό προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Europol, αλλά δεν έχει δώσει απαντήσεις λεπτομερέστερες στα ερωτήματά μας. Και πριν κλείσω θα ήθελα να πω ότι αυτές είναι οι απόψεις του των εκπροσώπων του Διοικητικού Συμβουλίου που λάβαμε γραπτός σε μια προκατακτική διαδικασία που ξεκίνησε όταν άρχισε η συζήτηση του θέματος αυτού. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ εγώ. Ε, πολύ μου άρεσε αυτό που αναφέρατε σχετικά με την Frontex. Να δούμε ο κύριος Φίντα Φάνινγκ, ο οποίος είναι ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠΟΛ. Να πάρει το λόγο παρακαλώ για να μοιραστεί τις ιδέες του μαζί μας. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Κυρίε και κύριοι, καλή σας μέρα. Η Αστυνομική Ακαδημία λαμβάνει ε, γνώση της ε, πρότασης ε, συγχώνευσης. Στην 29η ε, συνεδρίαση του το Διοικητικό Συμβούλιο ανέφερε τα εξής. Η συγχώνευση του ΣΥΠΟΛ και του ε, Europol δεν, ε, έχει, δεν είναι ευνοϊκή. Δεύτερον, θα πρέπει να υπάρχει εθνική συνεργασία με την Αστυνομική Ακαδημία, αλλά μέσω της συγχώνευσης αυτή η συνεργασία θα γίνει πιο δύσκολη. οι δομές των οργανώσεων, καθώς επίσης και τα υφιστάμενα δίκτυα σε επίπεδο ε, χωρών μελών παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές, κυρίως όσον αφορά τη διακυβέρνησή τους. Δεύτερον, η πρόταση θα σημάνει και μείωση ε, του διοικητικού προσωπικού που δεν μας φαίνεται πολύ ρεαλιστική θα πρέπει να καλύπτονται πάγιες ανάγκες και τώρα και στο μέλλον και επομένως δεν είναι λογικό να θεωρήσει κανείς ότι η Europol μέσω του προσωπικού της μπορεί να καλύπτει τις ανάγκες αυτές. Επιπροσθέτως, δεν έχει γίνει ε, ενδελεχής ε, υπολογισμός ε, από την Κομισιόν σχετικά με την χρήση του προσωπικού. Τρίτον, δεν ε, ε, είναι δυνατόν να υπάρξουν περαιτέρω ε, περικοπές και των δαπανών από την πλευρά της ΣΕΠΟΛ. Τέταρτον, η αύξηση των δαπανών και του κόστους για την κατάρτιση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να πω ότι μέχρι τώρα ε, μεγάλο μέρος των καταρτήσεων λαμβάνει χώρα ε, στις ε, χώρες μέλη που έρουν ένα σημαντικό μέρος του βάρους της κατάρτισης αυτής η οργάνωση τοπικών σεμιναρίων θα μπορούσε να διατηρηθεί μετά και τη συγχώνευση με την Europol. Πέμπτον, το γεγονός ότι η συνεργασία μεταξύ ε, Europol και Σεπολ λειτουργεί πάρα πολύ καλά είναι ακόμα ένα επιχείρημα κατά της συγχώνευσης. Υπάρχουν ε, πολλές ευρωπαϊκές ε, υπηρεσίες στην, στον τομέα της ασφάλειας ε, και μέχρι τώρα η καθεμία κάνει τη δουλειά της χωρίς επικαλύψεις η ε, ΣΕΠΟΛ έχει θέση ε, κατά της ε, συγχώνευσης μεταξύ της ΣΕΠΟΛ και της Europol και αναθέτει και στον παρόντα πρόεδρο αλλά και στους μελλοντικούς πρόεδρους να εκπροσωπεί την κοινή της αυτή θέση σε κάθε επίπεδο της διαδικασίας λήψης αποφάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή η απόφαση ελήφθη με ευρία πλειοψηφία τον Μάρτιο στην Διοικητική συνεδρίαση της ΕΣΕΠΟΛ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Σα ευχαριστώ εγώ. Θα ήθελα τώρα να ζητήσω τον κύριο ε, Μπάνφιλτ, ε, διευθυντή τη ΕΠΟΛ, να πάρει το λόγο. Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμοι βουλευτέ μέλη τη Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, κυρίε και κύριοι, θα ήθελα και εγώ να εκφράσω τι ευχαριστίες ε, μου που μα δίνει τη δυνατότητα να παρευρισκόμαστε σήμερα εδώ για να σα εκφράσουμε τις απόψει και του Διοικητικού Συμβουλίου της ε, Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας ε, που μου έδωσε και την εντολή να σας εκθέσω τις απόψεις τους. Βέβαια είναι δύσκολο να αποφύγουμε τις επαναλήψεις ε, γιατί οι δύο πλαίσαντες κύριοι έχουν στερήσει από μένα τα περισσότερα πυρομαχικά που είχα οπότε θα είμαι και σύντομος και θα προσπαθήσω απλά να συμπληρώσω τις δικές τους παρεμβάσεις. Όπως αναφέρθηκε λοιπόν τα τελευταία ε, δύο-τρία χρόνια, από το 2010 και μετά, η ΣΥΠΟΛ σημείωσε και αναγνώρισε την ανάγκη για αλλαγές. Και μετά το 2010 είμαστε στη φάση μίζωνας, μίζωνος αναδιάρθρωσης και στον τομέα της ε, διακυβέρνησης που είπατε. Μείωση σε μεγάλο ποσοστό είχαμε του κόστους διακυβέρνησης μειώθηκαν ε, οι συνεδριάσεις ε, του Διοικητικού ε, Συμβουλίου σε δύο, έγιναν κάποιες αναδιοργανώσεις επιτροπών ομάδων εργασίας και έτσι καταφέραμε να απλουστεύσουμε ακόμη περισσότερο την διακυβέρνηση. Το οργανισμό μας επίσης οι οικονομικοί πόροι που εξοικονομήσαμε διατέθηκαν για την ε, βελτίωση της αποδοτικότητας της ακαδημίας μας. Δηλαδή με σχετικά τον ίδιο ε, προϋπολογισμό από 2.000 ε, φτάσαμε σε 6.000 δράσεις και προσπαθούμε να χρησιμοποιούμε από το 2011 και μετά τεχνολογία εχμής τα έτη δηλαδή 2011 και 2012 ε, είχαμε πολύ περισσότερους ε, μάλιστα σπουδαστές ε, στα εικονικά μαθήματα, virtual μαθήματα που οργανώσαμε. Χρησιμοποιούμε και την κριτική προσέγγιση του Κοινοβουλίου και έχουμε βελτιώσει και τον τομέα της λογοδοσίας. Το 2012 κάναμε τον έκτο μας λογιστικό έλεγχο. Είμαστε ένας από τους οργανισμούς ε, με τους περισσότερους λογιστικούς ελέγχους, Θέλω να σας πω. Όλοι οι έλεγχοι δείχνουν ότι υπάρχει τακτικότητα, κανονικότητα και είμαστε και απόλυτα επιχειρησιακοί. Σε ό,τι αφορά τη βασική φιλοσοφία της ΕΠΟΛ, θέλουμε να βελτιώσουμε την συνεκτικότητά μας. Νομίζω ότι είμαστε πλήρως ενταγμένοι στο τοπίο το κοινοτικό σε ό,τι αφορά ε, την κατάρτιση που παρέχουμε. Η διδακτέα που προσφέρουμε πιστεύουμε ότι καλύπτει τις βασικές ανάγκες για την καταπολέμηση του σοβαρού οργανωμένου εγκλήματος. Συμμετείχαμε και στην ομάδα επαφής ε, δικαιοσύνης εσωτερικών. Θέλουμε μεγαλύτερο συντονισμό σε θέματα συντονισμού, και ε, μάλλον εκπαίδευση και κατάρτιση. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη συνεργασία μεταξύ Ευρωπόλ και ΣΥΠΟΛ, να σα πω δύο λόγια πάνω σε αυτό. Η ρήτρα συνεργασία δεν υπήρχε ποτέ, αλλά υπάρχει αυτή η συνεργασία τα τελευταία χρόνια και μπορείτε να βασιστείτε στην επαγγελματική συμβολή τη δική μας, όπως και εμείς βασιζόμαστε στην επαγγελματική συμβολή της ε, Ευρωπόλ για το περιεχόμενο, το χαρτοφυλάκιο των ε, μαθημάτων, ε, των εντοπισμών απειλών, για ένα νέο κύκλο πολιτικής που μπορούμε να προτείνουμε. Και έχουμε και 800 εκπαιδευτέ οι οποίοι ετησίως παρέχουν τα μαθήματα και η Europol προσφέρει 40 ειδικού εμπειρογνώμονες. Να σας πω όμως ότι οι εντολές των δύο αυτών οργανισμών δεν είναι οι ίδιες, διαφέρουν. 100 άτομα το φυλάκιο της ε, ΣΥΠΟΛ. Το 30% ασχολείται με θέματα που αφορούν το οργανωμένο εγκλήμα, ε, διασυναρικό έγκλημα. Και μιλάω για την κατάρτιση και το 70% έχει να κάνει με ανθρώπινα δικαιώματα, ε, ηγεσία, ε, διάφορες ε, κρίσεις, καταστάσεις εξανάγκης κτλ. Έχουμε μια συμφωνία σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο της εκπαίδευσης με την Ευρωπόλη. Θέλουμε να αντιμετωπίσουμε επιτυχώς ε, τις αυξανόμενες ανάγκες ε, εκπαίδευσης ε, στα όργανα επιβολής της νομοθεσίας, του νόμου. Μπορούμε να κάνουμε οικονομίες, αλλά πρέπει να σας πω ότι η επένδυση στην εκπαίδευση σημαίνει και επένδυση στην ασφάλεια. Σας ευχαριστώ πολύ και τώρα θα δώσω το λόγο στο Διευθυντή της Europol, τον κύριο Wainwright. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Καλημέρα, κυρίε και κύριοι. Όσον αφορά την πρόταση του κανονισμού, μερικέ πολύ γενικέ παρατηρήσει βεβαίω, θα γίνουν περισσότερε συζητήσει και ασφαλώ η Europol είναι έτοιμη να στηρίξει, να προσφέρει την αρρωγή της στην Επιτροπή στου επόμενους μήνες και ασφαλώς τον εισηγητή καθώς ετοιμάζει τη συζήτηση. Η Europol υποστηρίζει τις κύριες αρχές πίσω από την πρόταση, τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας στη λειτουργία και την λογοδοσία προς το Κοινοβούλιο, το υψηλότερο επίπεδο ε, παδοτικότητας και, και βέβαια την αποτελεσματική διακυβέρνηση. Και υπάρχουν πολύ σημαντικές και ενδιαφέρουσες προτάσεις ε, στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς την κατεύθυνση αυτή, ιδιαίτερα για τη βελτίωση της λειτουργικής αποτελεσματικότητας μιας υπηρεσίας η οποία αντιμετωπίζει έναν κίνδυνο πολύ πιο περίπλοκο, πιο δύσκολο για το οργανωμένο κυρίως έγκλημα από ό,τι έχουμε δει μέχρι τώρα και για την προστασία της, τις ε, ε, ασφαλιστικές δικλίδες για την προστασία. Εξετάζουμε με προσοχή τις προτάσεις, νέα στοιχεία και σημαντικές αλλαγές ως προς την συσχύουσες ε, ρυθμίσεις για την προστασία των δεδομένων της Europol που θα πρέπει βεβαίως να εξετάσουμε με προσοχή ώστε να μην περιοριστεί με την εισαγωγή αυτών α, μείωση στην αποτελεσματικότητα της λειτουργίας της ε, ε υπηρεσίας μας. Βεβαίως όλα αυτά με το πνεύμα συνεργαστείς με το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Για τη συγχώνευση με τη ΣΥΦΟΠΟΛ νομίζω ότι έχω πολύ, πολύ λιγότερο χώρο να προσθέσω σχόλια επιπλέον των όσων είπαν οι τρεις προλαλήσαντες. Ο Πρόεδρος μας είπε πολύ ξεκάθαρα ποιε είναι οι θέσει, δεν υπάρχει τόσο να αποκλίνω φυσικά από αυτό, αλλά αν μου επιτρέψετε θα προσθέσω κάποια τεχνικού χαρακτήρα στοιχεία στα, ε, στις παρατηρήσεις αυτές που σας μπορούν να, βοηθήσουν. Όπως είπε και ο Διευθυντής Μπάνφη, λοιπόν, μπορεί να υπάρξει ένα σύστημα κατάρτισης μέσα στη Europol. Μπορεί να υπάρξουν διαφορετικά μοντέλα και πρακτικές λύσεις για το πώς θα προσφερθεί αυτό. Δεν, αυ, δεν απαραίτητο δηλαδή, να περάσει μέσα από τη συγχώνευση τη Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία με την Europa, αλλά από την πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πάντω, αντιλαμβάνομαι ότι στόχο είναι κυρίω η βελτίωση τη αποτελεσματικότητα, την ε, κατάρτιση των αστυνομικών δυνάμεων και βέβαια έχει επιτελέσει υπάξια το έργο της ε, ΣΥΠΟΛ. Ε, Βεβαίω υπάρχει ένα πρόβλημα αντίληψης, κατανόησης των ζητημάτων της αστυνομικής συνεργασίας ακόμη, γιατί το βλέπω καθημερινά στη Europol, όπου πρέπει να ε, πείθουμε τους αστυνομικούς ε, από κάθε χώρα ότι υπάρχει ανάγκη και ότι είναι χρήσιμη η συνεργασία. Ακόμη και να έχουμε περάσει την κατάρτιση, υπάρχει ανάγκη λοιπόν για συνεργασία. Άρα το να έχουμε κάτι το οποίο μπορεί να δώσει μια καλύτερη ε, συνειδητοποίηση και κουλτούρα της συνεργασίας μεταξύ των αρχικών αρχών ασφαλώς και θα υποστηρίξουμε οποιαδήποτε τέτοια πρόταση. Επίσης συμφωνώ με τον ε, Διευθυντή Μπάνφη ότι συνεργάζονται πολύ ικανοποιητικά μεταξύ τους οι δύο ε, αρχές έχουν περίπου 30% ε, έχουμε περίπου το 30% των κοινών μαθημάτων που ανέφερε και ο κ. Μπάνφη. αν υπάρχει περιθώριο για περισσότερη συνεργασία τώρα. Εφόσον ληφθεί καταρχήν απόφαση για τη συγχώνευση, θα πρέπει και οι όροι αυτή τη συγχώνευσης να διατυπωθούν με μεγάλη προσοχή και κυρίως όσον αφορά τις επιπτώσεις του στη Europol, όπως άλλωστε ανέφερε μόλις τώρα ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ώστε να μην μετατραπεί σε ένα σημαντικό και νέο καθήκον για τη Europol ε, κατά τη στιγμή που δεν επαρκούν ε, ε, οι πόροι και οι ικανότητες της. Και πάλι για, το θέμα, για τα υπόλοιπα θέματα και εφόσον αποφασιστεί από την πολιτική εξουσία η συγχώνευση, θα πρέπει στην πράξη να αναζητήσουμε διαφορετικές λύσεις, όπως παραδείγματι θέματα χώρου ακόμα και για τα γραφεία μας, γιατί από τους υπολογισμούς που έχουμε τώρα μπορεί αυτό να καταστεί δυνατόν, αλλά οριακά ως προς τους χώρους γραφείων που διαθέτουμε αυτή τη στιγμή. Για να σας εξηγήσω συγκεκριμένα τι σημαίνει αυτό, έχουμε 865 θέσεις. Μπορούμε να χωρέσουμε στα γραφεία μας στη Χάγη 865. Αυτή τη στιγμή δουλεύουν 728 στο κτίριο αυτό, μαζί με κάποιες χειρεύουσες θέσεις που θα καλυφθούν και θα φτάσουμε κάπου στο 750-760 άτομα προσωπικού μέχρι το τέλος του χρόνου. Έτσι λοιπόν περισσεύουν το πολύ πολύ 60 γραφεία ή θέσεις γραφείου. Η πρόταση Ευρωπαϊκής προταση Ευρωπαϊκή προτείνει, μάλλον εκτιμά, τη δημιουργία νέων θέσεων 50 για το EC3 και άλλων 40 ε, για, το, για το τέταρτο τμήμα, τέταρτη υπηρεσία της Europol. Άρα ουσιαστικά καλύπτουμε, εξαντλούμε κάθε περιθώριο που έχουμε σε χώρο γραφείων. Και για να ολοκληρώσω θα παραλάβω αυτό που ακούσαμε και πιστεύω είναι το πιο σημαντικό στοιχείο από τόσο είπε ο Πρόεδρος μας στην παρέμβασή του ότι θα πρέπει να γίνει σεβαστή η ε, δυνατότητα της Europol να προσφέρει αποτελεσματική συνεργασία στα κράτη-μέλη. Εξαιρετώς τις αποφάσεις λοιπόν, που θα ληφθεί για τη συγχώνευση και για την αξιοποίηση των πόρων, δεν πρέπει να ξεχάσουμε ποιο είναι το βασικό μας καθήκον. Η συγχώνευση αυτή, εάν πρόκειται να γίνει, θα πρέπει να οδηγήσει σε καθαρό κέρδος για την ε, κοινωνία της επιβολής του νόμου και όχι σε επιδείνωση. Ευχαριστώ πολύ. Ε, θα δώσω τώρα το λόγο στους συναδέλφους βουλευτές. Ο κύριος Βάιντερ Χόρτερ θέλει το λόγο. Ναι, σιγά σιγά θα πάρετε όλοι. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με τους εγγραμμένους ομιλητές και θα δούμε. Ναι, Πρόεδρε, ευχαριστώ. Είναι κάπως ιδιάζουσα η συζήτηση που διεξάγεται εδώ. Έχουμε να κάνουμε αφενός με τη Europol και νομοθεσία η οποία έπρεπε από καιρό να έχει σαφθεί. Χαίρομαι ιδιαίτερος για την μεγάλη αισιοδοξία του εισηγητού που θεωρεί ότι θα μπορέσουμε να την ολοκληρώσουμε αυτή την προσπάθεια για την ομοθεσία, για το ομοθέτημα στην τρέχουσα θητεία. Είναι βέβαια πάρα πολύ σημαντικό για την Europol προκειμένου να προσφέρει την ευρωπαϊκή προσθέμενη αξία η Europol και ελπίζω ότι και οι πολίτες της Ευρώπης θα αναγνωρίσουν την ποιοτική δουλειά της Europol. Θα έχει λοιπόν την αναγνώριση και ως εκ τούτου και την ε, αντίληψη του πολίτη ότι προσφέρει κάτι θετικό στην Ευρώπη η Europol είναι κάτι πολύ θετικό και είναι πάρα πολύ σημαντικό βεβαίως να υπάγεται στον κοινοβουλευτικό έλεγχο, να λογοδοτεί στο Κοινοβούλιο η Europol. Αυτό είναι ένα θέμα πάρα πολύ σημαντικό. Επίσης πολύ σημαντικό για μένα είναι να δώσουμε ιδιαίτερη προστασία στις, ε, στην προστασία των προσωπικών δεδομένων. Ιδιαίτερα όσον αφορά την ε, ταυτοποίηση στοιχείων κατά τις έρευνες ε, που διεξάγονται και σε επίπεδο κρατών μελών, όλα αυτά σε ε, συνδυασμό με την όλη συζήτηση τη σχετική με το, με το σύνολο των μέτρων για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Πρέπει λοιπόν να μπορούμε να αποδώσουμε ε, να, να φέρουμε αποτελέσματα στην αστυνομική εργασία ταχύτατα και να συνεργάζεται και το Κοινοβούλιο με την Europol. Δεν καταλαβαίνω λοιπόν γιατί, παρότι είναι τόσο αργά για να το πω ευγενικά, στην θητεία μας ε, για να προχωρήσει αυτή η υπόθεση έρχονται ζητήματα προς συζήτηση τα οποία δεν έχουν κανένα λόγο να εμφανιστούν. Γιατί μπορούμε να μιλούμε βέβαια για συγχωνεύσεις, μπορούμε να μιλούμε για εξοικονόμηση πόρων. Αλλά είπατε και εσείς ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία η ε, προτεραιότητα που θα δοθεί στην ανεξαρτησία των ε, φορέων αυτών και ρωτώ, αφού έχουμε τόσο μεγάλη πίεση, γιατί ξαφνικά εμφανίζεται ένα νέο θέμα για να επιβαρύνει τη συζήτηση. Γιατί να δημιουργήσουμε ένα πρόβλημα το οποίο δεν θα έπρεπε καν να υπάρχει. Δεν θα ήταν καλύτερα να δούμε το ένα μετά το άλλο τα δύο αυτά νομοθετήματα και να αφήσουμε το ζήτημα της λειτουργίας ανοιχτό. Δεν βλέπω γιατί θα πρέπει σε τόσο ε, όψιμο στάδιο της θητείας μας να, να ανοίξουμε ένα τέτοιο κεφάλαιο. Ιδίω βέβαια δεδομένου ότι θέλουμε να κάνουμε ως το δυνατόν πιο γρήγορα τη δουλειά μας, που δεν πρέπει να χάσουμε το χρόνο μας. Ευχαριστώ η κυρία Ματιέ, μετά θα ακούσουμε και άλλους ομιλητές βεβαίως, αλλά θα ήθελα να παρακαλέσω να περιορίστε συνάδελφοι τις παρεμβάσεις σας στο 1,5 το πολύ λεπτό για να προλάβουν όσοι ενδιαφέρονται να λάβουν το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Λυπούμε που δεν ήμουν ε, από την αρχή των παρουσιάσεων. Όπως ε, ξέρετε, ε, ευθύνεται εν μέρη και σε μένα η πρόσκλησή τους. Εν πάση περιπτώσει, δυστυχώς ψηφίζαμε στην Επιτροπή Κρίμ για μια έκθεση η οποία είναι επίσης πάρα πολύ σημαντική. Σίγουρα θα μάθω τι είπατε, θα μου κάνουν μια σύνθεση. Η Ευρωπόλ βεβαίως ε, θα πρέπει οπωσδήποτε να είναι ανεξάρτητη γιατί κάνει ήδη πολύ σημαντική εργασία, κανείς δεν την αμφισβητεί και είναι μια εργασία πάρα πολύ ε, χρήσιμη για την ε, προστασία και την ασφάλεια των πολιτών γνωρίζουμε όλοι και το γνωρίζουν και όσοι εργάζονται στις δομές που μας απασχολούν σήμερα ότι η ασφάλεια των πολιτών είναι της ε, πρωτής του σημασίας ε, ε, βλέποντας τις εκθέσεις που μας κάνετε στα πλαίσια της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ διαπιστώνουμε ότι είναι δραματικά εντό εισαγωγικών τα στοιχεία και επομένως πρέπει να βελτιωθεί η κατάσταση. Κύριε Μπάνφη, από την άλλη μεριά ξέρουμε πολύ καλά την εργασία που κάνατε μετά από τις εκθέσεις της ΛΥΜΠΕ και της ΚΟΚΟΜΠΗ Πιστεύω λοιπόν και εγώ ότι αυτή η υπηρεσία θα πρέπει να παραμείνει ανεξάρτητη γιατί και η ΣΕΠΟΛΕ και η Ευρωπόλ έχουν λόγο ύπαρξης πρέπει να είναι ανεξάρτητες και να συνεργάζονται Καταλαβαίνω βεβαίω τι ανάγκες της Κομισιόν, καταλαβαίνω τις ανάγκες ε, για περιορισμούς ε, των ε, δαπανών. Πρόκειται για θέματα τα οποία όλοι γνωρίζουμε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις εθνικές δημοσιονομικές αρχές. Υπάρχει και μια πολιτική όσον αφορά την εκείνη την περιουσία. Και βεβαίως κατανοεί το μήνυμα της Κομισιόν το Κοινοβούλιο, αλλά ίσως θα πρέπει να βρούμε κάποιες άλλες λύσεις. Ξέρουμε ότι ο εισηγητής ε, ε, κύριος Δίας Δεμέρα είναι πολύ ανοιχτός. Είμαστε πολύ ανοιχτοί ε, να βρούμε λύση που θα ικανοποιεί και την Κομισιόν. Αλλά αυτή η πλήρης συγχώνευση δεν μας φαίνεται, δεν μου φαίνεται να είναι καλή ούτε για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή ούτε για τους Ευρωπαίους πολίτες, ούτε μακροπρόθεσμα για την κατάρτιση, την καλή κατάρτιση των των αστυνομικών στα 28 σε λίγο ε, κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, και μάλιστα αναφερόμενοι στην πρώτη μελέτη που είχε παραγγείλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτή η συγχώνευση φαίνεται να είναι η χειρότερη λύση γιατί μιλάμε για ανθρώπους ε, που ε, καταρτίζονται, εκπαιδεύονται για να διασφαλίσουν την ασφάλεια των πολιτών. Ελπίζω ότι εάν καθίσουμε όλοι γύρω από ένα τραπέζι και συζητήσουμε θα βρούμε κάποια λύση. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος, ε, η κυρία Χάνιστ. Ευχαριστώ. Πρέπει να διερωτηθούμε τι θέλουμε με αυτόν τον νέο κανονισμό της Europol. Μπορεί κανείς να κάνει, να επιχειρήσει τα πάντα, αλλά πρέπει να ξέρουμε τι θέλουμε. Πρέπει να είναι αποτελεσματική, διαφανής αστυνομική συνεργασία, αυτό είναι σίγουρο. Αυτό πρέπει να κάνουμε πάνω απ' όλο. Και αυτή είναι η πτυχή την οποία θα πρέπει να ερευνήσουμε αν θα ε, ικανοποιήσει, εξυπηρετήσει όποια συγχώνευση. Νομίζω ότι πρόκειται να το εξυπηρετήσει αυτό η συγχώνευση. Ή διαφορετικά λέμε δεν μας ενδιαφέρει η αστυνομική συνεργασία, περισσότερο μας ενδιαφέρουν τα ε, μέτρα αυτά κατάρτιση και μένουμε στο 30% που δεν είναι βέβαια ασφαλώς ο στόχος κανενός. Επίσης θα πρέπει να δούμε αυτό το black box. Θέλουμε η Europol να είναι ένα black box, ένα μαύρο κουτί που θα γίνει και μεγαλύτερο ακόμα με τη συγχώνευση. Γιατί εμείς ε, από την, ε, ομάδα, από την ΚΟΕ δεν επιδιώκουμε κάτι τέτοιο. Άρα δεν έχει κανένα λόγο να γίνει συγχώνευση. Εσείς αναφέρεστε βέβαια πάντα στον κανονισμό 2001, πολύ ωραία. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να κοιτάξουμε το πακέτο μέτρων για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, όπου δεν βλέπω καμιά προσπάθεια. Τέτοιου είδους κανονισμός λοιπόν για μένα δεν πρέπει, δεν χρειάζεται να εμφανιστεί σαν πρόταση όταν έχουμε το πακέτο για την ε, προστασία των προσωπικών δεδομένων, γιατί ασφαλώ θα την επηρεάσει. Η εκπρόσωπο τη Επιτροπή επίσης είπε ότι ε, θέλουν ε, οι εκθέσει να φτάνουν στα χέρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πάρα πολύ ωραία, καταπληκτικό. Αλλά τι σημαίνει αυτό συγκεκριμένα. Τι νόημα έχει δηλαδή, να τώρα που ξεκίνησε η συζήτηση με αυτόν τον κανονισμό και διαπιστώνουμε ότι η Europol είναι απολύτως αντίθετη με αυτή την ιδέα και την ε, διάθεση των ε, στοιχείων. Θα αλλάξουμε θέση σε αυτό ή όχι. Η διαφάνεια λοιπόν έχει πολύ μεγάλη σημασία και η προστασία των προσωπικών δεδομένων. Αυτό πάνω απ' όλα. Αυτά μέχρι τώρα. Σας ευχαριστούμε. Παρακαλώ πολύ κύριε Κίνγκ Νομίζω ότι όλες αυτές τις πληροφορίες που μας δώσατε ήταν πολύ σημαντικές. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντική η συνεργασία των αστυνομικών δυνάμεων στην Ευρώπη. Ε, ειδικά τώρα που γνωρίζει και ο κόσμος ποιες είναι οι δυνατότητες εργασίας σε επίπεδο επιβολής νόμου. Βεβαίως ε, η Europol χρειάζεται ε, πόρους για να ολοκληρώσει το έργο της. Αλλά εάν θέλουμε πραγματικά αποτελεσματική αστυνομική συνεργασία, προϋπόθεση απαραίτητη είναι η συνεργασία και η κατάρτιση. Έχουμε εδώ λοιπόν κάτι που από ό,τι έχουμε ακούσει λειτουργεί. Είναι καλό, είναι αποτελεσματικό. Επομένως δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να βρούμε κάτι άλλο, το οποίο όμως ε, είναι ασαφές γιατί δεν είναι 100% σίγουρο ότι θα δουλέψει ή θα λειτουργήσει καλά η συγχώνευση. Δεν νομίζω λοιπόν ότι η συγχώνευση θα ήταν καλή ιδέα. Συμφωνώ με τους προλαλήσαντες που είπαν ότι ενδεχομένως ε, είναι η χειρότερη δυνατή επιλογή. Εάν κάτι λειτουργεί, λειτουργεί καλά, έχει καλά αποτελέσματα, τότε πρέπει να το κρατήσουμε και να το ενθαρρύνουμε. Όχι να προσπαθήσουμε να του δημιουργήσουμε προβλήματα. Τη στιγμή που ήδη η λειτουργία του είναι τέτοια που λύνει προβλήματα. Ευχαριστώ πολύ. Δύο ακόμα εγγεγραμμένοι Σιλβί, Γκυγιόμ και ο Σλάβος Άλμπερτ και θα πω και εγώ δύο λόγια στο τέλος. Πολύ σύντομα κυρία Πρόεδρε γιατί τα περισσότερα έχουν ε, ήδη ε, υποθεί. Ε, ενδιαφέρουσα η συζήτηση πάντως ε, και στην τωρινή συζήτηση και στη, στα όσα μας είπε η Πρόεδρος του Κοινού Επιπτικού Οργάνου ε, ε, έχουμε την αίσθηση ότι όλοι μιλούν ελεύθερα και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Λοιπόν, για το θέμα της συγχώνευσης δεν το καταλαβαίνουμε. Σύμφωνα και με τις μελέτες που έγιναν, φαίνεται ότι τα πορίσματα είναι πάντα αρνητικά και επομένως δεν ξέρω, αναρωτιέμαι αν το, ο μόνος λόγος ε, και το μόνο κίνητρο είναι οικονομικό. Ε, δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να πάμε απευθεία στη συγχώνευση. Φαντάζομαι ότι μπορούν να βρεθούν ε, λύσεις οι οποίες θα αφορούν τη βέλτιστη χρήση των πόρων κτλ το μόνο ε, σημείο της ε, συγχώνευσης ίσως, ε, μάλλον όχι, από τη στιγμή που φαίνεται ότι είναι κόκκινο πανί το θέμα της συγχώνευσης θα πρέπει να δούμε πώς μπορεί να δομηθεί η συζήτηση, δηλαδή γύρω από ποια σημεία, που μπορούν να γίνουν εξοικονομήσεις, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικότερα τα χρήματα. Thank you very much, Chair, and... Άλμπερ, σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω και όλους σας ε, που είστε εδώ, όπως και η κυρία Ματιέ, στο συγγνώμη και εγώ που άργησα να έρθω, γιατί ψηφίζαμε στην ε, Επιτροπή ΚΡΙΜ την ενδιάμεση έκθεση. Και βέβαια πρέπει να σκεφτούμε και το μέλλον και του δικού μας εσωτερικού εδώ έργου για αυτά τα θέματα του οργανωμένου εγκλήματος ε, και του ελέγχου Πώ θα ασκεί τον έλεγχό της η Ευρωπόλ. Φυσικά και εμεί έχουμε τη θέση μας σε αυτή την όλη συζήτηση. Σε ό,τι αφορά πρώτα απ' όλα το ζήτημα της προστασίας δεδομένων, ε, σίγουρα είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του κανονισμού για την Ευρωπόλ και κατά την άποψή μου αν υπάρχουν ισχυροί κανόνες προστασίας δεδομένων, αποκτά μεγαλύτερη εξοπιστία η Ευρωπόλ. Ιδίω αν βλέπουμε ότι υπάρχει ισχυρότερη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αστυνομικών αρχών. Άρα ε, έντονη είναι και ανάγκη για μεγαλύτερη προστασία των δεδομένων. Άρα και η οδηγία για την προστασία των δεδομένων είναι σημαντική στον τομέα της επιβολής του νόμου. Πραγματικά λοιπόν απευθύνω έκκληση σε όλους σας αλλά και σε όλους εμάς να επιμείνετε τα κράτη-μέλη να συμφωνήσουν ε, επί μιας δέσμης κοινών κανόνων. Αυτό κατά την άποψή μου αποτελεί προϋπόθεση. Έτσι το βλέπουμε ως κοιόδης. Ως προϋπόθεση. Δηλαδή να προσαρμοστεί η οδηγία αυτή και μετά να ενισχύσουμε και την ανταλλαγή πληροφοριών στο πλαίσιο της Ευρωπολ, γιατί οι αστυνομικέ αρχές σε όλα τα κράτη-μέλη θα πρέπει να μπορούν να εμπιστεύονται τα συστήματα των άλλων κρατών μελών. Επομένως, τις δεσμευτικούς, τους δεσμευτικούς αυτούς κανόνες, κοινούς κανόνες τους χρειαζόμαστε. Ας εργαστούμε από κοινού όλοι λοιπόν και α εξετάσουμε αυτά τα ζητήματα από κοινού. Αυτό αποτελεί προπόθεση και νομίζω το χρειαζόμαστε. Από πλευρά Κοινοβουλίου θα επιμείνουμε. Και αν μου επιτρέπετε μια τελευταία φράση, και συγγνώμη που μακρηγορώ, για τη ΣΥΠΟΛ και τη συγχώνευση. Συμφωνώ απόλυτα με αυτό που είπαν οι συνάδελφοι. Η ανεξάρτητη αστυνομική ακαδημία έχει την αξία της. Και επίσης, ό,τι αφορά την ενίσχυση της Ευρωπόλ στον τομέα και του προϋπολογισμού, θέλω να πω ότι και αυτό είναι προτεραιότητα. Είναι προτεραιότητα στον προπολογισμό μας. Και αν προχωρήσουμε και δαπανίσουμε εκατοντάδες εκατομμύρια για UPNR ή για τα εφή e σύνορα. Φυσικά και θα μείνουν λιγότεροι πόροι για την καλή δουλειά που κάνουν οι κοινέ ερευνητικέ ομάδε τη Europol. Αυτά όλα θα τα συζητήσουμε και όταν θα συζητήσουμε τον προλογισμό μα. Ευχαριστώ. Η Πρόεδρο, αν με επιτρέπετε να προσθέσω και εγώ κάποια σχόλια. Βλέπετε εδώ ότι έχουμε δύο ε, οργανισμούς που λειτουργούν πολύ καλά. Και έχουμε μια πρόταση πολύ σημαντική για όλους μας. Και πρέπει το συντομότερο δυνατόν να καταλήξουμε πριν το τέλος της κοινοβουλευτικής αυτής περίοδου. Όμως εδώ βλέπουμε ότι η όλη αυτή η ιδέα της συγχώνευσης μας δυσκολεύει τη δουλειά. Είναι μια πρόταση που δεν είχε ε, προετοιμαστεί τόσο καλά. Δεν άκουσα να μιλήσει κανείς υπέρ της συγχώνευσης. το μόνο επιχείρημα είναι η ενδεχόμενη εξοικονόμηση κάποιων πόρων και δεν είναι και κάτι που μας έχει πείσει. Σίγουρα είναι ανάγκη να εξοικονομούμε πόρους, αλλά δεν μας έχει πείσει ότι θα γίνει αυτό σε συγκεκριμένη περίπτωση. Πρέπει να προχωρήσουμε λοιπόν με αυτή την νομοθετική πρόταση στο συντομότερο δυνατόν, η οποία περιλαμβάνει σημαντικά ε, στοιχεία, προστασία δεδομένων, πώς θα γίνει πιο επιχειρησιακή η Europol. Θα ήθελα να συνεχίσουμε τη συζήτηση αυτή και ακούστηκαν πιστεύω πολύ ε, σημαντικά επιχειρήματα. Θα ήθελα να ακούσω τα καταληκτικά σχόλια του εισηγητή μας του κυρίου Ντίαφ Ντεμέρα. Παρακαλώ. Τα τελικά σας σχόλια. Ντίαφ Ντεμέρα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Πράγματι εκτιμώ όλος ιδιαιτέρως τις ε, παρουσιάσεις ε, που ακούσαμε από τη ΣΥΠΟΛ και την Europol και από τους ε, πρόεδρους των διοικητικών συμβουλίων και από την πλευρά των παρουσιάσεων των διευθυντών τους. Μετά λοιπόν από όσα άκουσα, πού καταλήγω. Βλέπω ότι έχουμε μία δέσμη επιχειρημάτων που είναι κατά της συγχώνευσης. Τα περισσότερα επιχειρήματα είναι νομίζω εύλογα και μπορούμε να τα συνοψίσουμε ως εξή. Η αποτελεσματικότητα των δύο οργάνων είναι κάτι που μπορούμε να πιστοποιήσουμε και φυσικά ότι χρειάζεται να βελτιωθεί ακόμη περισσότερο και αυτό το προσυπογράφουμε. Λογικό είναι επίσης ότι εάν λειτουργούν με ένα λογικό τρόπο χωριστά αυτές οι δύο υπηρεσίες, γιατί να μπούμε σε περιπέτειες συγχώνευσης που είναι και αβέβαιο το μέλλον και η επιτυχία της ε, άσκησης αυτής. Δεν φαίνονται συμπαγή τα επιχειρήματα υπέρ αυτής της πρότασης. Ούτε ως προς την ε, κατεύθυνση εξοικονόμησης πόρων, δεν είναι βέβαιο αυτό, ούτε είναι βάσιμο το επιχείρημα ότι θα βελτιωθεί με τον τρόπο αυτό ο συντονισμός η συνεργασία των δύο αυτών υπηρεσιών, που μέχρι στιγμή λειτουργεί πολύ καλά. Είναι λοιπόν ε, αμφισβητήσιμη η εφαρμογή του άρθρου 88, το είπα και εγώ. Πρέπει να βρεθεί λοιπόν ένα πιο λογικό νομικό επιχείρημα και να μην επικαλούμαστε μόνο το άρθρο 88 επειδή απλά και μόνο κάνει λόγο για ε, την εκπαίδευση. Ως καθήκον. Εκτιμώ λοιπόν πάρα πολύ και τη διάθεση όλων να συνεργαστούν με την Επιτροπή. Ο Διευθυντής της Ευρωπόλη επίση είπε ότι είναι διαθέσιμος να ε, οργανώσει στο δυνατόν όλες τις απαιτούμενες άτυπες συναντήσεις. μετά από την ανάλυση και τα σχόλια των ε, συναδέλφων επίσης, για την επόμενη άνοιξη, ε, επειδή το Μπράνσιλ τέλειωσε, μας τέλειωσε, έτσι είπαν οι Βρετανοί, ε, σταματάμε, πρέπει να βρούμε λοιπόν, πρέπει να δούμε τι πιστεύουμε, είμαστε κατά, όπως από ό,τι φαίνεται είμαστε, τη συγχώνευση και αν ναι, πρέπει να βρούμε ένα νέο Μπράνσιλ. Αυτό γιατί το λέω. Γιατί ο Ρομπ Βάινράιτ ολοκληρώνοντας την παρέμβασή του, είπε ότι ένα από τα προβλήματα στη Χάγη είναι το πρόβλημα του χώρου. Πρέπει να το σκεφτούμε αυτό. Θέλω να ευχαριστήσω πραγματικά ε, πολύ θερμά τους συναδέλφους από την ε, Σοσιαλιστική Ομάδα αλλά και από το ΕΛΚ αλλά και από τις άλλες ομάδες. Τα σοσιαλδημοκρατικά σχόλια ήταν πολύ ευπρόσδεκτα. Πράγματι, αχρίαστα περιπλέκουμε τη ζωή μας και τα πράγματα με ε, το να ασχολούμαστε με αυτό το θέμα της συγχώνευσης. Συμφωνώ απόλυτα με τη Βερονίκ Ματιέ. Δεν μου φαίνεται καλή ιδέα η πλήρης ε, η ολική συγχώνευση. Μπορεί να πρέπει να εξετάσουμε άλλα ενδεχόμενα. Δεν μου φαίνεται καλή ιδέα της συγχώνευσης για την κυρία Ένστα η οποία διερωτάται αν έχει λόγο ύπαρξη σε συγχώνευση. Αυτό το συζητούμε. Και επίσης οι Χέρμς και Άλμπρεχτ επίσης έχουν εκφράσει την ίδια ανησυχία δηλαδή όλα τα θέματα τα οποία ε, τον της προστασία των δεδομένων και είναι στον κανονισμό Ευρωπόλ θα πρέπει να μπουν στο ευρύτερο αυτό φάσμα το οποίο συζητούμε στο Κοινοβούλιο. Οδηγία σας δεδομένων για το οποίο θέμα είναι αρμόδιος ο συζήτης ο κ. Άλμπρεχτ. Κίνγκα Γκάλ. Μιλήσατε για τη σημασία της αστυνομικής συνεργασίας στην Ευρώπη. Και επισημάνατε κάτι που είναι προφανές. Αν λειτουργεί η συνεργασία, γιατί πρέπει να αλλάξει, δεν πρέπει. Και ολοκληρώνω με τον Αντιπρόεδρο. Ε, συμφωνώ και εγώ ότι ε, είναι πολύπλοκο το θέμα της ε, συγχώνευσης. Και δεν ακούστηκε εδώ κανένα επιχείρημα που να συνηγορεί πέρα αυτής. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε πώς θα προχωρήσουμε στον τομέα αυτό τη προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μην ξεχνώντα όμω ότι έχουμε και να κάνουμε έναν οργανισμό που ασχολείται με την ασφάλεια. Αυτά είχα να πω. Σα ευχαριστώ πολύ όλου για τι παρεμβάσει σα, γιατί πραγματικά εμπλούτησαν και τη δική μου σκέψη και θα μείνω πολύ χρήσιμη. ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ όλους όσους συμμετείχαν σε αυτήν την μακρά συζήτηση, αλλά θα συνεχίσει η δουλειά πάνω στην νομοθετική πρόταση. Λοιπόν, έχουμε ακόμα ένα σημείο στην διάταξη. Λοιπόν, θα σας αποχαιρετήσουμε και μετά θα συνεχίσουμε τη συνεδρίασή μας. Ε, Όπως είπα και προηγουμένως, έχουμε ακόμα ένα σημείο στη μέση διάταξή μας. Πρόκειται για τη συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Τουρκίας για την επενιστοχή προσώπων που διαμένουν χωρίς άδεια. Η συγγήτρια η κυρία Ζόμερ και παρακαλώ τη Ρενάτε να λάβει το λόγο για να μας παρουσιάσει συνοπτικά Τι συστάσεις της. Και ο κύριος Λουτσάνο Φραντσέσκο είναι εδώ, από τη, ενημερώνομαι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ευχαριστώ όλους όσοι έλαβαν μέρος στην προηγούμενη συζήτηση. Κυρία Ζώμερ. Κοιτάξτε, όποιο δεν συμμετέχει στο επόμενο θέμα στη συζήτηση, παρακαλώ τις συζητήσεις του να τις δεξάγει στο διάδρομο. Αφήστε εμάς που θέλουμε να δουλέψουμε στο τελευταίο σημείο της ημερής διάταξη. Κυρία Ζώμερα, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να αναφερθώ και να παρουσιάσω σήμερα την έκθεση για την επανεισδοχή προσώπων, χωρίς ε, συγκεκριμένο όμως χρονοδιάγραμμα της σχέση με την Τουρκία. Έχουμε βέβαια και τις ε, προθεσμίες για τις τροπολογίες ε, και τις δικές μας προθεσμίες ανεξάρτητα από την υπογραφή της επανεισδοχής από την ίδια την Τουρκία αλλά κάποια στιγμή πρέπει και εμείς να ασχοληθούμε με το θέμα αυτό και χαίρομαι που ήρθε η ώρα να το συστήσουμε σήμερα. Τι έχουμε λοιπόν. Το Νοέμβριο του 2002 ήδη η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Τουρκία συμφώνησαν την ε, σύναψη μιας ε, συμφωνίας για την επανεισδοχή των παρανόμως διαμενόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση προσώπων. Πέρασαν 8 χρόνια και στις 14 Ιανουαρίου του 2011 ολοκληρώθηκαν αυτές οι διαπραγματεύσεις και τον Ιούνιο του 2012 έγινε η μονογραφή της συμφωνίας. Απαιτείται η σύμπραξη του Κοινοβουλίου στη διαδικασία αυτή. Είναι μια συμφωνία πάρα πολύ σημαντική για την Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι όλοι γνωρίζουμε ότι οι οδοί, οι μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας είναι αυτές που αποτελούν και την κύρια, που, που, από την οποία περνάει η κύρια ροή των παρανόμων μεταναστών ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ως εκ τούτου απαιτείται να προχωρήσει η συμφωνία της επανεισδοχής που σημαίνει ότι η χώρα από την οποία έχουν ε, μπει τελευταία στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι παράνομοι μετανάστες ε, επαναπροωθούνται στη χώρα προελεύσεως τους. Η Τουρκία μέχρι τώρα μόνο έχει μονογράψει τη συμφωνία. Προϋπόθεση για την υπογραφή της συμφωνίας καθιστά την κατεργασία ενός προγράμματος, ε, ενός φίλου πορείας για την απελευθέρωση από τα καθεστώς του διαβατηρίου από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εν τέλει ε, δεχόμενη αυτή την απέτηση της Τουρκίας καταθέτει μία πρόταση, ένα πρόγραμμα δράσεως συγκεκριμένα για την απελευθέρωση της θεωρούς των διαβατήριων με πολύ αυστηρά κριτήρια ωστόσο. Ε, απαιτεί δηλαδή νομοθετικές και διοικητικές μεταρρυθμίσεις από πλευράς της Τουρκίας σε σχέση με την ε, διασφάλιση των εγγράφων ταυτότητας και την διαφύλαξη των θεμελιωδών ε, δικαιωμάτων, όλα αυτά σε σχέση με την απελευθέρωση της υποχρέωσης θεώρησης διαβατηρίων. Η Συμφωνία Επανεισδοχής για την Ευρωπαϊκή Ένωση βεβαίως έχει μεγάλη σημασία, όπως είπα. Είναι σημαντική συμβολή στην ε, χαλιναγώγηση της παράνομης μετανάστευσης. Ταυτόχρονα μπορεί και να βοηθήσει τον έλεγχο και καταπολέμηση της υπερσυνοριακής εγκληματικότητας, δεν έχουμε να κάνουμε διακίνηση ανθρώπων κυρίως, και να αποφορτήσει από αυτό το βάρος αντίστοιχα την Ελλάδα που είναι κρατός μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ως εκ τούτου και την Ευρωπαϊκή Ένωση γενικότερα στο ζήτημα της ρύθμισης και ε, του ελέγχου της νόμιμης μετανάστευσης. Ως εκ τούτου το πρόγραμμα δράσης για την σταδιακή απελευθέρωση θεώρηση των διαβατήριων από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί ένα βήμα προς τις προϋποθέσεις, προς τις επιθυμίες της Τουρκίας και πιστεύουμε και ότι και η Τουρκία θα πρέπει να κάνει από πλευρά της το καθήκον της. Από πλευρά Τουρκία τώρα, η κύρωση τη διαδικασία αυτή, συμφωνία αυτή, φαίνεται να προγραμματίζεται ώστε να καθυστερήσει τόσο μέχρι ότου προσφερθεί από πλευρά Ευρωπαϊκή Ένωση η απελευθέρωση από τη θεώρηση διαβατηρίων από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για του Τούρκου υπηκόου, πράγμα το οποίο κρίνω απαράδεκτο. Άλλωστε, στην τελευταία έκθεση πρόοδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καταγράφεται και υπογραμμίζεται ξεκάθαρα ότι η Τουρκία θα πρέπει να κάνει σεβαστή την ε, ε, ακαιρεότητα τη Ευρωπαϊκής Ένωση, στο σύνολό τη πράγμα το οποίο δεν γίνεται επουδενή, άλλωστε το αποδεικνύει και η ε, στάση η αρνητική, η απορριπτική που είχε έναντι της Προεδρίας της Κυπριακής Δημοκρατίας στο δεύτερο εξάμεινο του 2012 για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν έχει αναγνωρίσει ω ανεξάρτητο κάτω την Κυπριακή Δημοκρατία η Τουρκία και πρέπει να πούμε και να το καθιστούμε καθημερινά σαφές ότι με τον τρόπο αυτόν παραβιάζει, δεν αναγνωρίζει στην ακαιρεότητά της, το ολόκληρό της, το όλον της, την Ευρωπαϊκή Ένωση Τουρκία. Η Τουρκία επίσης ε, δεν πληρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το πρωτόκολλο, το προσεκτημένο συμφωνία σύνδεσης ε, έναντι της Κύπρου. Δηλαδή δεν πληρεί τις ε, υποχρεώσεις που απορρέουν έναντι του συνόλου των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης η έκθεση προόδου επίσης υπογραμμίζει αυτά τα στοιχεία και σημειώνει ε, προβλήματα και ως προς την ελευθερία της έκφρασης, τις θεμελιώδεις ελευθερίες και δικαιώματα, τα προβλήματα στη λειτουργία της δικαιοσύνης, την ελευθερία της θρησκευτική συνείδησης, όλα αυτά τα οποία δεν συνάδουν με τις ευρωπαϊκές αρχές και αξίες. Η Τουρκία μέχρι τώρα δεν έχει πληρεώσει σε κανένα σημείο τα πολιτικά κριτήρια της Κοπεχάγης και ως εκ τούτου είναι πάρα πολύ σημαντικό να το επισημάνουμε και εν ώψη της συζήτησης για τη Συμφωνία Επανεισδοχής, γιατί όλα αυτά ε, έρχονται σε αντίθεση με τις ε, διαπιστώσεις της εκθέσεως προόδου ε, για τις εξελίξεις στη χώρα αυτή και τον πολιτικό διάλογο με την Ευρωπαϊκή Ένωση εν όλο. Και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό και σωστό η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή πλευρά, στο πρόγραμμα δράσεως για την απελευθέρωση των ε, θεωρήσεων να διατηρήσει τις ε, υψηλές προδιαγραφές, τα αυστηρά κριτήρια τα οποία έχει θεσπίσει και η τουρκική πλευρά παρά τις ε, υποχωρήσεις και παραχωρήσεις που έχουμε κάνει προς το πρόγραμμα δράσης για την θεώρηση των διαβατηρίων έχει δείξει ακόμη παρελκυστική πολιτική, καθυστερεί ακόμη περισσότερο, προσπαθεί να μας επιβάλλει πιέσεις προκειμένου να χορηγηθεί πρώτα η απελευθέρωση της θεωρής νηβατηρίων και μετά να κινηθεί η τουρκική πλευρά, πράγμα το οποίο βρίσκω εγώ δυσανάλογα ε, δυσανάλογη συμπεριφορά. Θα έπρεπε η Τουρκία να εκπληρώσει το δικό της μερίδιο των υποχρεώσεων και να δώσει ένα θετικό μήνυμα ε, προς την Ευρωπαϊκή Ένωση εν ώψη αυτής της συμφωνίας για την επανεισδοχή. Είναι κάτι από το οποίο θα επωφεληθεί όχι μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και η Τουρκία ίδια η συμφωνία επανεισδοχής ανοίγει το δρόμο εν τέλει στην απελευθέρωση της θεωρίας των πατηρίων και εν όλο βοηθάει την προσέγγιση της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Τουρκία με τη συμφωνία αυτή εξάλλου θα υποφεληθεί και από την οικονομική και τεχνολογική υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ε, ανάπτυξη και την κατάρτιση της, ε, του σώματος συνοριοφυλάκων και τεχνική υποστήριξη της τη των συνόρων. Σημαντικό επίσης είναι να σημειώσουμε ότι μέχρι τη θέση σε εφαρμογή και την ουσιαστική λειτουργία της ε, συμφωνίας, οι εκρεμείς διμερείς συμφωνίες έναντι των κρατών με τα οποία έχετε τη συμφωνία στην Τουρκία θα πρέπει να εφαρμόζεται κατά τρόπο συσταλτικό. Και θα ήθελα να ρωτήσω εάν αυτή η συμφωνία αν είναι δυνατόν να υλοποιηθεί, τι είδους επιπτώσεις θα έχει στις διμερείς συμφωνίες σε σχέση με τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία ε, Τουρκία έχει καθυστερήσει εδώ και τέσσερα χρόνια την υλοποίηση των συμφωνιών αυτών. Και ζητώ από το Συμβούλιο να λάβει μια σαφή τοποθέτηση της Τουρκίας και να καλέσει την Τουρκία άνευ χρονοτριβής να υλοποιήσει, να ε, κυρώσει, να υπογράψει και να κυρώσει και να υλοποιήσει χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση τη Συμφωνία Επενδυτικής. Και όπως είπα και στην αρχή, όσο δεν έχει υπογράψει τη συμφωνία αυτή η Τουρκία, ούτε εμεί μπορούμε να δώσουμε την έγκρισή μας για τη συμφωνία από πλευράς Ευρωπαϊκής. Ούτε μπορούμε να συμφωνήσουμε στην ε, υπόθεση αυτή μέχρι ότου η Τουρκία δείξει διάθεση για συνεργασία. Μέχρι τότε θα περιμένουμε. Νομίζω ότι αυτή ήταν μια πάρα πολύ σαφής παρουσίαση ενός αμφιλεγόμενου ζητήματος. Ε, η σημασία που αποδίδουν οι συνάδελφοι στο θέμα αυτό αποδεικνύεται από τον μακρύ κατάλογο αγοριτών. Εφτά είναι οι συνάδελφοι οι οποίοι θέλουν να πάρουν το λόγο. Να σας πω ότι θα ήθελα να σας ε, ζητήσω μονάχα ένα λεπτό να μιλήσετε ο καθένας. Ε, κυρία Μποσκούρ πρώτα απ' όλα. Ένα λεπτάκι και θα μου δώσετε τη δυνατότητα σας παρακαλώ να σας πω πότε πέρασε το ένα λεπτό. Ε, θα είμαι πάρα πολύ σύντομη. Γιατί η συγγήτρια είπε πολλά και θα ήθελα να αντιδράσω. Ε, e Μιλάμε για συμφωνίες επανεισδοχής ε, ε, προσώπων, ε, αλλά κάθε φορά που έχουμε περάσει τέτοια συμφωνία, αυτομάτως υπάρχει και άρση της υποχρέωσης ε, θεώρησης για τους πολίτες της εν λόγω χώρας. Αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι έχουμε ήδη συμφωνίες επανεισδοχής που λειτουργούν. Δεν θέλουμε να υπάρχουν συμφωνίες χωρίς αντίκρισμα γιατί αυτό θα σημαίνει περισσότερα προβλήματα από όσα αντιμετωπίζουμε ήδη λόγω της ε, λαθρομετανάστευσης. Νομίζω ότι και η Ελλάδα έχει ήδη ε, συμφωνία επανεισδοχής που αντιμετωπίζει όμως πολλά προβλήματα. Το είδα άλλωστε και σε μια επίσκεψη εργασίας που είχα κάνει στην Ελλάδα πριν από ένα χρόνο πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι το αποτέλεσμα θα είναι καλό και για τις δύο πλευρές, γιατί διαφορετικά δεν πρέπει να λειτουργήσει το σύστημα θα πρέπει η συμφωνία επανεισδοχή να είναι επωφελής ε, για όλους, έτσι ώστε και για τα δύο μέρη, έτσι ώστε να τη δεχτούν βλέποντας την παρούσα κατάσταση στην ε, ε, Τουρκία υπάρχουν πέντε κέντρα υποδοχής χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση που όμως αποτελούν αντικείμενο αντιδράσεων από μη κυβερνητικέ οργανώσεις οι οποίες δεν είναι αρκετά. Τέλος πάντων θα πρέπει να συζητηθεί, να μελετηθεί το θέμα περισσότερο ε, εάν θέλουμε πραγματικά να λειτουργήσει ε, το σύστημα επανεισδοχής. Ούτως ή άλλως το παρόν σύστημα δεν επιτρέπει την πραγματική λύση του προβλήματος γιατί ε, ξαναφεύγουν αυτοί οι παράνομοι μετανάστες προς τις χώρες. επίσης Υπάρχουν κάποιες ακραίες καταστάσεις που αντιμετωπίζει η Τουρκία αυτή τη στιγμή, π.χ. στα σύνορα με τη Συρία. Να υπογραμμίσω ότι το, υπάρχει το μνημόνιο κατανόησης το οποίο έχει υπογραφεί μεταξύ Frontex και Τουρκίας και αυτό είναι θετικό. Ήδη δημιουργείται μια κοινή έτσι, διαδικασία συνεργασία κοινός πολιτισμός συνεργασία με την Τουρκία. Και ένα τελευταίο, οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις φοβούνται ότι ενδεχομένως θα χρησιμοποιηθεί η ε, συμφωνία επανεισδοχής έτσι ώστε να απομακρυνθούν από ευρωπαϊκές χώρες ε, Τούρκοι εργαζόμενοι οι οποίοι δεν είχαν το χρόνο τη δυνατότητα να ανανεώσουν την άδεια παραμονής εργασίας τους εκεί. Εν ολίγης λοιπόν θέλουμε να υπογραφεί η Συμφωνία Επανεισδοχής, αλλά θέλουμε ταυτόχρονα να λύσουμε και τα προβλήματα. Ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόεδρος. Η ε, κυρία Γκρισπέκ. για ένα λεπτό όμως εσείς, αν είναι δυνατόν. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Πάρα πολύ σύντομα. Και εγώ θέλω να πω ότι επί της αρχής δέχομαι, στηρίζω την προσέγγιση της εισηγητρίας, αλλά ε, δεν στηρίζομαι ε, όλη την επιχειρηματολογία της ή τον τρόπο που αυτή ε, δομείται σε σχέση με την Συμφωνία Δοχής. Έχω και μία ε, και ένα σχόλιο πολιτικό, έχω μια, ένα σχόλιο που κάνω συνήθως, αυτό είναι το εξής. Η Κομισιόν μας έχει δώσει ε, διαρκώς πληροφορίες σχετικά με τις συμφωνίες επανεισδοχής που έχουν ολοκληρωθεί και που, έχουν, που βρίσκονται ε, ε, υποσυζήτηση, αλλά θεωρώ ότι δεν μας έχει δώσει πολλές πληροφορίες όσον αφορά την επανεισδοχή ας πούμε ατόμων βάσει της συμφωνίας με το Πακιστάν το 2010. Η ασφάλεια των προσώπων αυτών μας ανησυχεί ακόμα. Γι' αυτό λοιπόν ε, θέτω διαρκώς αυτήν την ε, ερώτηση, γιατί ξέρετε δεν είναι ε, υπογράφω μια συμφωνία επανεισδοχής, επαναπροωθώ τους ανθρώπους και τελείωση. τελείωσε. Έχω επίσης και μια ανησυχία να εκφράσω. βλέπω ότι παρουσιάζονται ε, κάποιες ελλείψεις ε, όσον αφορά την οργάνωση της ε, χώρας στην Τουρκία, ελευθεροτυπία, ελευθερία των μέσων ενημέρωσης, ανεξαρτησία της δικαστικής εξουσίας, ας πούμε η Ρεπόρτερ χωρίς σύνορα λένε ότι η Τουρκία είναι η μεγαλύτερη φυλακή για τους δημοσιογράφους. Επομένως είναι πάρα πολύ σημαντικό να τα ξαναδούμε αυτά. Είναι πολύ σημαντικό να δούμε και το ζήτημα των ε, ε, θεωρήσεων ε, ταξιδίου. Η βίζα φυσικά είναι ένα σημαντικό θέμα που πρέπει να λυθεί και μεταξύ της Τουρκίας και της Ευρώπης γιατί αυτή τη στιγμή είναι η μόνη υποψήφια χώρα ε, η οποία δεν έχει δει απελευθέρωση ε, του συστήματος των θεωρήσεων ενώ υπάρχουν χώρες οι οποίες ε, όπως η Μολδαβία η Ουκρανία δεν χρειάζονται πλέον βίζα και που δεν είναι και υποψήφιες. Ε, θα πρέπει λοιπόν ε, να μπορέσουμε να απελευθερώσουμε, να ανοίξουμε το δρόμο έτσι ώστε στον ευρωπαϊκό χώρο να έχουμε και ανταλλαγή απόψεων, ερευνητών κτλ. Και άλλα θα είχα να δεν έχουμε το χρόνο. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. 20 λεπτά είχε ε, προβλεφθεί για τη συζήτηση αυτού του περιπλόκου ζητήματος. Κυρία Ένστ, παρακαλώ, για ένα λεπτό. Ναι, τρία σημεία. Κυρία Ζόμερ. Τι θέλετε δηλαδή. Θέλετε να συνάψετε μια συμφωνία με ένα κράτος το οποίο από ό,τι πολύ σωστά επικρίνεται δεν τηρεί τα συμπεφωνηθέντα και από την άλλη διαμαρτύρεστε που δεν κάνει η Τουρκία αυτά πρέπει να κάνει. Αυτό ενώ από την άλλη την ε, θεώρηση των διαβατηρίων την έχουμε δώσει σαν απελευθέρωση ως δώρο λίγο πολύ στα κράτη τα οποία είναι στα πρόθυρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για όλα τα κράτη αυτό έγινε. Γιατί να μην θέλει και η Τουρκία την απελευθέρωση. Δηλαδή θα πρέπει να συνάψει συμφωνία η Τουρκία, την οποία όμως δεν θέλει αυτή τη στιγμή να συνάψει, την οποία δεν έχει καν κυρώσει όταν καλά-καλά δεν ξέρουμε τι περί τίνος πρόκειται. Και επίσης πρέπει να πούμε ότι δεν είναι ακριβώς η κοιτίδα της δημοκρατίας η Τουρκία. Ας μην είμαστε ε, υπερβολικοί. Υπάρχουν πάρα πολλές ε, παραβιάσεις των ανθρωπινών δικαιωμάτων. Ας ξεκινήσω με τους Κούρδους βεβαίως, αλλά και πολλά άλλα ζητήματα, στα οποία είναι, είμαστε επικριτικοί, όπως και για την Κύπρο βεβαίως. Και γι' αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε ποιος, ποιον αφορά όλο αυτό το πράγμα. Έχουμε να κάνουμε με την ε, Συρία, με εκατοντάδες χιλιάδες Σύρων ε, προσφύγων, πολλές χιλιάδες ε, απατρίδων, μεταναστών κτλ. που υποτίθεται ότι βρίσκονται στην Τουρκία και τους οποίους θα πρέπει να επαναδεχθεί η Τουρκία. Στην ε, Γερμανία με επίσημα στοιχεία 10.000 ήταν ε, οι υποψήφοι προς επαναπροώθηση. Άρα λοιπόν νομίζω ότι πριν να συστήσουμε κάτι τέτοιο θα πρέπει να προσκαλέσουμε την υπατιαρμοστία των Ηνωμένων Εθνών ε, για τα ανθρώπινα δικαιώματα, να συζητήσουμε ξεκάθαρα τα θέματα αυτά, να έχουμε μια σαφή εικόνα και μετά να κάνουμε προτάσεις για ε, ε, σύναψη συμφωνίας, κύρωση κτλ. Να έχουμε πρώτα μια σαφή εικόνα. Ευχαριστώ πολύ. Έχω ακόμα τον κύριο Κλέης, παρακαλώ αλλά προσπαθήστε να μην ξεπεράσετε το ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ορθώς η εισηγήτρια μας λέει ότι η Τουρκία είναι ε, η κύρια χώρα από την οποία περνάει το μεγαλύτερο μέρος της λαθρέας μετανάστευσης. Ε, επομένως πρέπει να υπάρξει, συμφωνία, να υπάρξει συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Τουρκίας. Είναι γεγονός ότι υπήρξε μέγα πολιτικό σφάλμα από πλευρά των Ευρωπαϊκών ε, της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης ε, να συνδέσει την Συμφωνία Επενεισδοχής με τη Συμφωνία για τις Θεωρήσεις. Μέγα σφάλμα. Το κάναμε, το σφάλμα αυτό και με άλλες χώρες, αλλά η Τουρκία είναι μια ειδική περίπτωση, λαμβάνοντας υπόψη τις, τους τεράστιους αριθμούς παρανόμων μεταναστών που περνούν από την Τουρκία. Η Τουρκία εκβιάζει αυτή τη στιγμή αρνούμενη την συμφωνία επανεισδοχής μέχρι ότου υπάρξει συμφωνία για την κατάργηση της βίζας. Θα πρέπει να αντισταθούμε σε αυτήν την στάση, γιατί διαφορετικά θα αντιμετωπίσουμε εκ νέου μια κατάσταση κατά την οποία δεν θα γίνονται σεβαστοί οι κανόνες. Δηλαδή η Τουρκία ε, θα καταφέρει να ε, έχει επιτύχει ε, την κατάργηση της θεώρησης, δεν θα χρειάζεται πλέον βίζα, αλλά από την άλλη μεριά δεν θα σεβαστεί την Συμφωνία Επανεισδοχής. Δηλαδή από τη μία πλευρά προσπαθούμε να μειώσουμε την παράνομη μετανάστευση μέσω της Συμφωνίας Επανεισδοχής, από την άλλη ανοίγουμε τις πόρτες διάπλητες σε παραπάνω μετανάστευση με την άρση της θεώρησης. Κύριε Φλότ, για ένα λεπτό. Α, δεν είναι πολύ ένα λεπτό. Είμαι και πρόεδρος αντιπροσωπείας με την Τουρκία. Θέλω λίγο περισσότερο χρόνο. Είναι πολύπλοκη συζήτηση και βλέπουμε ότι αυτά τα οποία είπε η κυρία Ζόμερ για την κατάσταση στην Τουρκία ε, ουσιαστικά μια έκθεση πρόοδο για την Τουρκία και όλες οι φαντασιώσεις περί ε, μετανάστευσης ε, υπάρχουν στην συζήτηση αυτή και τελικά κάνουν ακόμα πιο θολό το ήδη ε, πολύπλοκο αυτό ζήτημα. Και ο Διευθυντή Frontex μα είπε ότι το ζήτημα της διέλευση ε, διαχερσαίων συνόρων Ελλάδας-Τουρκίας δεν είναι πλέον ε, το κύριο ζήτημα, ότι έχουν αλλάξει οι διαδρομές, είναι μέσω Βουλγαρίας ε, ή διαθαλάσσης. Άρα ήδη αυτές τις δεν θίγουμε σωστά το θέμα στη συζήτηση. Έπειτα, ε, το πολιτικό momentum. Είναι και αυτό ένα θέμα. Εσείς ε, θα αναλάβετε την υποχρέωση ε, και θα πιέσετε τώρα την Τουρκία όταν πραγματικά είναι τόσο μικρές οι δυνατότητες υποδοχής σύρων προσφύγων στην Ευρώπη και όταν η Τουρκία μόνη της 400.000 σύρους πρόσφυγες υποδέχεται. Πιστεύετε ότι είναι σωστή επιλογή πολιτική στιγμής να πούμε στην ε, Τουρκία να δεχθεί Σύρους πρόσφυγες ε, που θα φτάσουν παρά τους φραγμούς που βάζουμε εμείς στο ευρωπαϊκό έδαφος. έχω ε, νομίζω ότι υπάρχουν κάποια όρια στην πολιτική λογική και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη. Αυτό το momentum δεν είναι το κατάλληλο, κατά την άποψή μου, για να συζητήσουμε τη συμφωνία πανεζακής με την Τουρκία. Δεύτερον, Υπάρχει συζήτηση που επανέρχεται και ξανά επανέρχεται για τις ε, συμφωνίες επανεισδοχής. Αυτή που διαπραγματευτήκαμε με την Τουρκία ε, είναι μια συμφωνία που δεν ε, είναι καθόλου βελτιωμένη σε σχέση με την πρόταση της Κομισιόν και η ίδια η Κομισιόν είχε πει ότι είναι λίγο αμφίβολο το κατά πόσον μπορούμε να αξιολογήσουμε και να έχουμε μια συνέχεια ε, με τους ε, επαναπροωθούμενους. Ελάχιστες είναι οι βελτιώσεις, ελάχιστα είναι τα νέα στοιχεία που μάλλον θα ε, ενθαρρύνουν τις παραβιάσεις των ε, κανόνων, αφού δεν χρειάζεται διαβατήριο απλά ένα λεσέ πασέ και με μια μαρτυρία μπορεί να γίνει. Έχουμε μια επιτροπή επανεισδοχής που θα έχει την πλήρη αρμοδιότητα, αδιαφανέστατα όλα αυτά και εμείς δεν έχουμε και μέσα να ασκήσουμε ως κοινοβούλιο τον ε, δημοκρατικό κοινοβουλευτικό έλεγχο. Και όσον αφορά το ίδιο το αντικείμενο είναι πολύπλοκο. Και για να ολοκληρώσω, Προσθέτω και το γεγονός ότι η Τουρκία από αυτή την πλευρά υφίσταται και μία άνηση μεταχείριση. Κάτι πολύ επιζήμιο σε αφορά τη δική μας ε, εικόνα στην Τουρκία, όταν αυτή τη στιγμή εγκρίνεται και ένας νέος για τους πρόσφυγες, όταν η Τουρκία ζητά βοήθεια από την Ευρώπη για τον έλεγχο και τη συγκράτηση των ε, μεταναστευτικών ορών και για το σεβασμό των δικαιωμάτων ε, των μεταναστών. Σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση την προενταξιακή εκφράζει κάποιες ανησυχίες ε, για τη χρηματοδότηση των πέντε κέντρων κράτησης αντί να στηρίζονται οικονομικά οι μεταρρυθμίσεις ε, στο ποινικό δικαστικό σύστημα και στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Υπάρχουν ζητήματα λοιπόν, διακόπτη πρόεδρος. Εντάξει, ολοκλήρωσα. Σημαντικά πάντως όλα αυτά τα θέματα και πρέπει να τα λάβουμε υπόψη μας. Yeah. Το μικρόφωνο της Προέδρου έχει κλείσει. Λοιπόν, γνωρίζουμε, καταλαβαίνουμε ότι ο προβλεπόμενος χρόνος συζήτησης είναι πολύ λίγος για ένα τόσο σημαντικό ε, ζήτημα, αλλά βεβαίως ε, ε, δεν έχουμε περισσότερο χρόνο. Ο κύριος Τριανταφυλλίδης, παρακαλώ, για ένα λεπτό αν μπορείτε κι εσείς. Thank you, Chair. I won't take more than one... Ευχαριστώ πολύ. Δεν θα ξεπεράσω το ένα λεπτό, δεν θα επαναλάβω αυτά που είπαν άλλοι συνάδελφοι. Αλλά θα ήθελα να ε, συγχαρώ την εισηγήτρια κυρία ε, Σόμερ, γιατί έθιξε πολλά ε, ανοιχτά ζητήματα, κυρίως όσον αφορά την συμπεριφορά της Τουρκίας απέναντι στην Ευρώπη. Ανέφερε ορθώς η κυρία Ζόμερ ότι η Τουρκία δεν έχει καν σεβαστεί την εδαφική ακαιρεότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στα πλαίσια και της ε, Κυπριακής Προεδρίας εάν δεν σέβεται την ε, ε, Κυπριακή Προεδρία θα δεχτεί ας πούμε τη συμφωνία για όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή για 27 πλήν της Τουρκίας, πλήν της Κύπρου. Ε, ε, επίσης υπάρχει το ζήτημα ε, των κατεχομένων εδαφών γιατί ξέρετε μπαίνουν στα κατεχόμενα οι παράνομοι μετανάστες περνούν την πράσινη γραμμή και επομένως βρίσκονται σε ευρωπαϊκό έδαφος. Ευχαριστώ πολύ. κυρία Καλέρη είναι η τελευταία ομιλήτρια. Σας ευχαριστώ. Θα προλάβω κι εγώ ότι για την απελευθέρωση από τη θεώρηση των διαβατηρίων είναι κάτι το δεδομένο. Δεν θα έπρεπε ένα κράτος ε, μέλος να έχει υποχρέωση ε, θεώρησης. Θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε λοιπόν ταχύτερο δυνατό να ε, ελαφρύνουμε αυτή την υποχρέωση. Και η θέση του διαβατηρίου πάντοτε ήταν ε, να μην μιλάει για παράνομους μετανάστες, γιατί δεν υπάρχει κανένας άνθρωπος που είναι παράνομος, αλλά για παράτυπη μετανάστευση. Αυτή είναι η σωστή ορολογία. Θα ήθελα επίσης να επισημάνω ότι δεν μιλούμε την έκθεση πρόοδου της Τουρκίας, αλλά ε, μια συμφωνία επανεισδοχής και γι' αυτό το λόγο δεν χρειάζεται να αναφερόμαστε σε διάφορα άλλα ζητήματα όταν έχουμε μάλιστα πολύ σημαντικές προόδους καταγράψει και για τη μεταρρύθμιση του δικαστικού και για το κουρδικό ζήτημα, καλό είναι να μην αναφέρονται μόνο τα αρνητικά. Και θα ήθελα να ρωτήσω το εξή. Εάν είναι τόσο φρικτή η κατάσταση στην Τουρκία, γιατί θέλουμε να επαναπροωθήσουμε εκεί ανθρώπου που έρχονται να ζητήσουν άσυλο και προστασία. Δεν καταλαβαίνω, εφόσον δεν τηρείται καμία ε, αρχή και αξία. Είναι πολύ σημαντικό, ωστόσο, το δικαίωμα στο άσυλο, το σύστημα του ασύλου, ε, το οποίο στην Τουρκία βελτιώνεται σχετικά με τη νέα νομοθεσία για τη μετανάστευση, αλλά δεν υπάρχει επαρκής ακόμη νομοθεσία για τους ετούντε στο άσυλο. Γιατί λοιπόν να μην υπογράψουμε εμείς τη Συμφωνία Επανεισδοχής. Ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόεδρος, και θα ήθελα να παρακαλέσω την κυρία Ζόμερ να μας κάνει μια πολύ σύντομη ε, συνοπτική απάντηση στα θέματα αυτά. ασφαλώ δεν είναι τελευταία φορά που συζητάμε το θέμα. Είναι πολύ περίπλοκο και δύσκολο. Σας παρακαλώ να είστε στο δυνατόν πιο σύντομοι για να προχωρήσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Πάρα πολύ σύντομα. Ως εισηγήτρια, εδώ μόνο την αιτιολόγηση και το υπόβαθρο μπορώ να παρουσιάσω και γι' αυτό ε, προσπαθώ να εξηγήσω γιατί χρειάζεται αυτή η συμφωνία επανεισδοχής. Η θέσεις που εκφράζονται πολλές φορές όμως στην, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι πολύ έντονες και θεωρώ ότι η προσβλητική και η βριστική έκφραση, οι ανοησίες που είπε η κυρία Πρόεδρος της Επιτροπής ε, ή της Αντιπροσωπείας για τη σχέση με την Τουρκία, η κυρία Φλότρο, για τα λόγια μου, ο χαρακτηρισμός αυτός είναι απαράδεκτος και τον επιστρέφω. Οτιδήποτε άλλο έχετε να πείτε, συζητήστε το καλά, δεν υπάρχει λόγος να ξεφτελιζόμαστε έτσι. Ε, για τη συμφωνία λοιπόν αυτή εμείς μπορούμε να πούμε μόνο ναι ή όχι. Αν θέλετε να καταθέσετε τροπολογίες, η μόνη τροπολογία που μπορούσατε να καταθέσετε θα ήταν η απόρριψη ή η αποχή. Τίποτα περισσότερο δεν μπορείτε να πράξετε. Και θα ήθελα επίσης ε, να σημειώσω ότι έχουμε να κάνουμε με, με υπογραφή από πλευρά μα, δηλαδή έγκριση ή απόρριψη. Τίποτε άλλο δεν έχουμε να διαπραγματευτούμε, να τροποποιήσουμε. Σα ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόεδρο. Λυπούμε γιατί θα πρέπει να κλείσουμε πάνω σε αυτήν νότα διαφωνίας δεν μπορώ να κάνω τίποτα άλλο. Ένα σημείο μόνο έχει μείνει η προστασία των φυσικών προσώπων ενάντια τη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τι αρμόδιε αρχέ για το σκοπό τη πρόληψη, τη διερεύνηση, τη διαπίστωση ή τη δίωξη αξιόπινων πράξεων ή τη εκτέλεση ποινικών κυρώσεων και ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών. Δεν διαβάζω όλο τον τίτλο. Και συζητούμε το θέμα αυτό του κυρίου Δρούτσα. Παρακαλώ λοιπόν τον εισηγητή να συνοψίσει και να δώσει τις ε, προτάσεις του για τους συναδέλφους και την Επιτροπή που είναι εδώ παρούσα. Θα είναι θαύμα αν καταφέρετε μέσα σε 10-15 λεπτά να ολοκληρώσουμε το θέμα. Παρακαλώ. Ε, Ευχαριστώ πολύ. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομος κύριε, κυρία Πρόεδρε για να μην χάσουμε πολύ χρόνο. Πρώτα απ' όλα, στο συγγνώμη τη ζήτησα αναβολή της συζήτησης ε, Ξέρετε ότι έχουμε μια προσέγγιση δέσμης, ε, δηλαδή οδηγία και κανονισμός μαζί, αλλά επειδή γιορτάζαμε το Ορθόδοξο Πάσχα, ε, είναι μια πολύ σημαντική θρησκευτική ότι για εμάς ε, ζήτησε την αναβολή και σας ευχαριστώ πολύ που τη δεχθήκατε. Πολύ σύντομα λοιπόν θα ήθελα να σας ενημερώσω για το ότι οι συναντήσεις μεταξύ σκιωδών βαίνουν ομαλώς. Ήδη έχουμε συζητήσει έναν αρκετά μεγάλο όγκο, ε, ένα μεγάλο μέρος της οδηγίας. Συνεχίζονται οι εργασίες ε, των σχεδόν και ξέρετε ότι η προτεραιότητα και ο στόχος μας είναι η ευθυγράμμιση της οδηγίας με τον κανονισμό για την προστασία των δεδομένων. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο χρειάστηκε να συντονίσουμε τις εργασίες μας με τις συναντήσεις των σκιωδών για τον κανονισμό, διότι μπορούν αυτά τα αποτελέσματα ενδεχομένως να ενσωματωθούν και στις συζητήσεις για, τον, για την οδηγία. Με τον Γιάνν Άλμπρεχτ πάντως και τους άλλους αδέλφους η συνεργασία μας είναι άψογη. Στο πλαίσιο αυτό να πω ότι καταβάλουμε προσπάθειες ε, για να καταλήξουμε σε συμβαστικές τροπολογίες και λαμβάνουμε υπόψη μας και τη συμβολή, τις συστάσεις ε, του επόπτη για την προστασία δεδομένων και επίσης το, την ομάδα εργασίας για το άρθρο 29. Έχω ενημερώσει και τον Γιάννα Αλμπρέχτ ε, και πρέπει να σας πω και σε εσά ότι δεν πρέπει να υποτιμούμε ότι πρόκειται για πολύ μεγάλο όγκο δουλειά και μάλλον φαίνεται πρακτικά ανέφικτο να καταφέρουμε να έχουμε ολοκληρώσει τις εργασίες με βάση την προθεσμία που ορίσαμε. Ευθύ εξ αρχή είχαμε πει ότι είναι πάρα πολύ φιλόδοξο ο στόχο αυτό. Θέλαμε η ψηφοφορία στην Επιτροπή μα ε, να λάβει χώρα περί τα τέλη Μαου, Ήδη ο Γιάννα Αλμπρεχτ χθε είπε ότι δεν φαίνεται να είναι εφικτό κάτι τέτοιο και θα πρέπει να αναβληθεί η ψηφοφορία. Εμεί θα κάνουμε πάντω κάθε προσπάθεια να επιταχύνουμε τη δουλειά μα και να την ολοκληρώσουμε το συντομότερο δυνατό ώστε να μπορέσουμε να ψηφίσουμε πριν τι θερινέ διακοπέ. Αυτή είναι μια ε, δυνατότητα. Μπορούμε ίσω να έχουμε ολοκληρώσει μέχρι το καλοκαίρι. Και αν μου επιτρέπετε για ένα ακόμα λεπτό κυρία Πρόεδρε, να αναφερθώ στο άκρο προσφυλές μα συζήτημα τη οδηγία για την προστασία των δεδομένων τη λεγόμενη προσέγγιση πακέτο. Ξέρετε ότι ενοχλώ ε, τους συναδέλφους ε, με όλες τις δηλώσεις ε, και παρεμβάσεις μου για αυτό το θέμα και θα το επαναλάβω δυστυχώς για μια ακόμη φορά διότι και πάλι ε, κυκλοφορούν φήμες και ίσως είναι και κάτι περισσότερο από αυτό για το ότι τελικά φαίνεται να υπάρχει ε, μία ε, μειοψηφία εμπλοκή στο ε, Βούλιο. Δηλαδή, ο δημόσιο τομέα θέλουν να εξαιρεθεί και να περιληφθεί στην οδηγία ο δημόσιο τομέα, να εξαιρεθεί από τον κανονισμό. Ο κύριο Νίμιτ, φαντάζομαι θα επαναλάβει σήμερα τα ίδια, είχε επισημάνει ότι αυτό θα υποβαθμίσει ε, τα επίπεδα προστασίας που χαίρουν σήμερα, των οποίων χαίρουν σήμερα οι πολίτες μας, δυνάμει της προηγούμενης οδηγίας. Αυτό θα πρέπει να το λέμε πολύ σοβαρά υπόψη μας ως ε, κοινοβούλιο. Και να ενημερώσω τους συναδέλφους για το εξής. Στη συνάντηση των σκιωδών συζητήσαμε και αποφασίσαμε, γιατί ξέρετε υπάρχει μια μεγάλη ποικιλία νομικών μέσων στον τομέα ε, της επιβολής του νόμου και του ποινικού δικαίου. Πρέπει να έχουμε ή δυνατόν ένα κοινοτικό πρότυπο, ένα κοινωνικό κανόνα για την προσέγγιση των δεδομένων. Έχουμε διάφορες διαδικασίες που ε, είναι σε εξέλιξη. Έχουμε αυτή τη συμφωνία για το EUPNR που συζητείται αυτή τη στιγμή. Έχουμε το πακέτο για την ε, νομιμοποίηση των ε, προσόδων από παράνομε δραστηριότητε, το ξέπλυμα χρήματο, δηλαδή, το πακέτο για την Ευρωπόλ επίσης. Περιμένουμε το λάβουμε εδώ στο Κοινοβούλιο σύντομα, άρα υπάρχει αυτή η έντονη ε, αλληλεπίδραση και διαλειτουργικότητα μεταξύ αυτών και των σχετικών με την προστασία των δεδομένων διατάξεων. Κατόπιν κοινή συμφωνία λοιπόν των σκιωδών εισηγητών έστειλα επιστολή στον πρόεδρο και τους συντενιστές της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ ζητώντας τους να εξετάσουν το ενδεχόμενο την έγκριση ορισμένων ε, των μέσων που σας προανέφερα να συνδεθεί με την πρόοδο ή και την έγκριση ενδεχομένως της οδηγίας. Νομίζω ότι ως Κοινοβούλιο και από πολιτικής πλευράς θα πρέπει να εξετάσουμε τον ενδεχόμενο αυτό για να στείλουμε ένα απαραίτητο μήνυμα στους συναδέλφους ε, στο Συμβούλιο, συναδέλφους από κάποια κράτη-μέλη. Και το λέω και ανοιχτά να ασκήσουμε και την απαιτούμενη πίεση. Πρώτα, σε ευχαριστώ πολύ. Να δούμε ποιος θέλει το λόγο. Α, ο Γιάννα Άλμπρεχτ, που είναι ο συγκητής. Ποιος άλλος θα ήθελε να πάρει το λόγο. Ωραία, καταγράφω τους αγορητές. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο κύριος Άβλερτ. Ευχαριστώ πολύ και τον Δημήτριο Δρούτσα για την εξαιρετική εργασία του. Τώρα προσπαθούμε να συνεργαστούμε έτσι ώστε να ε, ευθυγραμμιστούμε κατά κάποιο τρόπο. Ε, και βεβαίως ε, η δουλειά μας ε, δείχνει ότι είναι δυνατόν να έχουμε καλά αποτελέσματα. Και θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι περιμένουμε και από τους άλλους συνομοθέτες μία αντίστοιχη στάση. Επίσης βλέπουμε ότι υπάρχουν ε, διασυνδέσεις σημαντικές ε, θέλουμε να ευθυγραμμιστούμε όσον αφορά ορισμούς και θέσεις των δύο ε, των δύο εγγράφων. Ε, υπάρχουν ορισμοί όσον αφορά τα, τον χαρακτηρισμό των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που δεν είναι ε, σαφής. Ε, λαμβάνοντας υπόψη και την προηγούμενη συζήτηση με τη Europol είναι σαφές ότι χρειαζόμαστε κοινά ε, στοιχεία, κοινή ε, αντιμετώπιση των πληροφοριών, του τρόπου ανταλλαγής ε, πληροφοριών. Χρειαζόμαστε εμπιστοσύνη ε, και αμοιβαία δέσμευση. Γι' αυτό λοιπόν είμαι βέβαιος ότι θα μπορέσουμε να λύσουμε τα προβλήματα τα οποία έχουν προκύψει Νομίζω λοιπόν ότι και στις ερχόμενες εβδομάδες θα καταφέρουμε να συνεργαστούμε ακόμα καλύτερα και θα τελειώσουμε αυτά τα δύο θέματα γρήγορα. Ναι, είναι, είναι ε, τεράστια δουλειά. Κορνίλια Έρνστα. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς ευχαριστώ θερμά τον εισηγητή. Και θα ήθελα να πω ότι εδώ έχουμε έναν πολύ σοβαρό, ένα πολύ σοβαρό θέμα να λήξουμε, αν βρισκόμαστε σε ισότιμη θέση με το Συμβούλιο ή όχι, να μην βρισκόμαστε δηλαδή σε αυτήν την ε, σφαλμένη τροχιά ε, που ε, μας προσπαθεί να μας βάλει το Συμβούλιο. Και εδώ νομίζω ο κύριος Τρούτσες το έχει πολύ ξεκάθαρα πει. Το θέμα αυτό των θεμελιδών ελευθεριών βεβαίως έχει ε, διατυπωθεί, έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε το Κοινοβούλιο να έχει μια γενική τοποθέτηση και μόνο εδώ με το πακέτο για τις ε, και την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μπορούμε να τοποθετηθούμε εμείς πιο ξεκάθαρα. Σημαντικό είναι να είναι συμβατό, όπως είπε και ο προλαλής σας. Μιλήσαμε νωρίτερα για την Europol, όλα αυτά πράγματα ε, ε, που βλέπουμε να συμβαίνουν ουσιαστικά αποτελούν ε, μια παραβίαση, δεν είναι συμβατά δηλαδή με τις βασικές αρχές. Και γι' αυτό θα ήθελα το Συμβούλιο να δείξει ειλικρινή στάση. Διαφορετικά δεν έχει νόημα να ε, παλεύουμε με τις σκιές. Ελπίζω, λέει πρόεδρο, να παλεύουμε μόνο με σκιέ. Σα ακούσουμε το Συμβούλιο και την Προεδρία. Ο κύριο Νέμιτ είναι εδώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, πρόεδρε. Η δική μα αξιολόγηση είναι αντίστοιχη με αυτή του εισηγητού. Σημειώνουμε καλή πρόοδο σε επίπεδο Συμβουλίου και στο Κοινοβούλιο. Πιστεύουμε ότι μπορεί να οδηγήσει σε καλά αποτελέσματα. Προτείνουμε βεβαίως ένα πακέτο το οποίο θέλουμε να προχωρήσει. Ένα πακέτο με δύο νομοθετήματα. Για δε το θέμα της δημοσίας τάξεως δεν νομίζω ότι έχουν κλείσει συζητήσει. Ε, πρέπει καταρχάς να συζητήσουμε και να ξεκαθαρίσουμε τι εννοούμε. Ε, γιατί η συνθήκη λέει ότι τα μέτρα τα σχετικά με, την, ε, με τον νόμο και την τάξη είναι στα χέρια των κρατών μελών. Από την άλλη πρέπει να υπάρχει και η συνένεση ότι δεν θέλουμε να ε, όπιστοδρομήσουμε σε σχέση με τις υφιστάμενες προδιαγραφές προστασίας και εφαρμογής του νόμου σε σχέση με τα ε, σήμερα ισχύονται. ισχύοντα. Όλα αυτά λοιπόν κινδυνεύουν να μας πάνε πολύ πίσω. Γι' αυτό οι αντιπροσωπείες οι οποίες τώρα έχουν ξεκινήσει αυτή τη συζήτηση για τα θέματα της δημόσιας τάξης, καλό θα ήταν να ξεκαθαρίσουν τι εννοούν. Νομίζω ότι ουσιαστικά είναι πολύ κοντά σε μια θέση αντίστοιχη με το άρθρο 72. Δεν βλέπω ανασχετική ε, πλειοψηφία η πρόταση για μεταφορά όλων των προτάσεων στην οδηγία. Δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να ζητήσει κάτι τέτοιο ε, χωρίς και να εκτεθεί στις κατηγορίες ότι υποβαθμίζουμε σοβαρά τις προδιαγραφές που είχε ορίσει η οδηγία του 95. Κάθε άλλη πρόταση βέβαια είναι ευπρόσδεκτη και ε, θετική. με, την, ε, με το σύστημα της συνθήκης ε, έχουμε κάνει την πρόταση για τα δύο νομοθετήματα γιατί έχουμε διαφορετικά κεφάλαια που καλούνται από διαφορετικά νομοθετήματα και θέλουμε να διαφυλάξουμε το σύστημα της συνθήκης, δηλαδή οδηγία πλαίσιο για το ποινικό ε, σκέλος και τις σχετικές δραστηριότητες και γι' αυτό προτείνουμε και την οδηγία. Μία λογική η οποία δεν θα ίσχυε σε περίπτωση που μεταφέραμε θέματα από το ένα στο άλλο. Άρα λοιπόν, για να μην ακυρωθεί, να μην αναιρεθεί το πνεύμα της συνθήκης, έχει κάνει την πρόταση για τα δύο νομοθετήματα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό θεώρησα καλό να το επισημάνω, γιατί δεν θα ήταν σκόπιμο να δημιουργηθεί, να δοθεί εντύπωση ότι υπάρχει μια τάση έντονη προς την κατεύθυνση αυτή. Έγιναν κάποιες διερευνητικές προτάσεις, αλλά νομίζω ότι μπορούμε με βάση την πρόταση της ε, ε, επίτροπή να δώσουμε λύσεις που θα βελτιώνουν σε σχέση με τα ισχύοντα εδώ και 10 χρόνια στο τομέα αυτών. Ε, βεβαίως, όπως είπατε, θα πρέπει οι ουσιώδεις κανόνες να απασχολήσουν τα άλλα θεσμικά όργανα, αλλά είπατε και εσείς ότι υπάρχουν και άλλες. Ε, η Πρόεδρος ε, ενημερώνει ότι σταματούν οι διερμηνείς. Να είστε σύντομος, γιατί θα φύγουν οι διερμηνείς. Ναι, Πρόεδρε, ε, η ουσία των αποφάσεων για την προστασία των δεδομένων και οι προτάσεις που κάναμε για τεχνικούς λόγους δεν επεκτείνονται. Αλλά αυτό ακριβώς έχουμε πει από την αρχή στην πρότασή μας. Ευχαριστώ πολύ. Καλώς λέει ο Πρόεδρος. Λίγα σύντομα σχόλια λοιπόν από την Προεδρία